Ε, ευχαριστώ. Σίγουρα η διάσκεψη της Νέας Υόρκης ε, ε, στη διάσκεψη αυτή μάλλον συμμετείχε μέλη αντιπροσωπεία και από το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την σύντομη επισκόπηση που μας κάνατε του έργου της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης. Είναι σημαντικό να μιλούμε για την επανεγκατάσταση σε συνδυασμό με την ένταξη και φυσικά ανάγκη ενίσχυση της επανεγκατάστασης. Επιπλέον, ας μην ξεχνούμε ότι ε, τη μερίδα της ευθύνης την αναλαμβάνουν κυρίως φτωχότερες χώρες, αλλά υπάρχει πολιτική και ανθρωπιστική ε, ευθύνη και υποχρέωση και, των Ηνωμένων, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και φαίνεται ότι και οι χώρες αυτές θα κληθούν να αυξήσουν τους αριθμούς προσφύγων που λαμβάνουν προς επαναγκατάσταση. Είμαι σαφώς και εγώ και η ομάδα μου υπέρ της επαναγκατάστασης σε συνδυασμό με την ένταξη. Βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο. Και μερικές φορές γίνονται έως και σπασμωδικές ιστερικές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Ε, και το γεγονό ότι ε, θα πρέπει να ξεχνούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από τις αντοχές της κοινωνίας μας. Ε, δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς ε, με την πείρα σας, την πλούσια και την εμπειρογνωμοσύνη σας ε, να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας για να ε, περάσουμε το μήνυμα ότι όχι μόνο θα πρέπει να επαυτούσουμε τις προσπάθειές μας για να προστατεύσουμε τους πλέον ευάλωτους, αλλά και να περάσουμε το μήνυμα ότι μόνο έτσι θα αντισταθμίσουμε ή θα βάλουμε το αντίβαρο σχέση με τα αρνητικά μηνύματα δυστυχώς που κυκλοφορούν. Ο Κάρλος, ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε την εμπειρία σας και τις γνώσεις για το θέμα αυτό. Συμφωνώ καταρχήν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα επιμέρους δεν έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν αυτό τον καταιγισμό προσφύγων και αυτό είχε αφενός σχέση με την ανθρωπιστική κρίση που έλαβε χώρα στη Μεσόγειο, αλλά επειδή δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τα αίτια του προβλήματος, στη ρίζα του. Από ό,τι κατάλαβα από την ομιλία σας, ε, πιστεύετε κι εσείς και συμφωνώ μαζί σας ότι η επανεγκατάσταση είναι ε, από τους πιο ασφαλείς διάβλους για την υποδοχή προσφύγων και είπατε περιλημμένως ότι ε, θα πρέπει να δεχτούμε πάνω από 500.000 ε, ε, πρόσφυγες για επανεγκατάσταση την επόμενη πενταετία. Μήπως είναι συντηρητική αυτή η εκτίμηση. Δεν θεωρείτε ότι παρά είναι συντηρητική. Κύριε κυρία Μπιόρκη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Μίλιμπαν που είχε την καλοσύνη να έρθει και ευχαριστώ και τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης που εκπροσωπεί για το τεράστιο έργο και τη συμβολή της στον τομέα αυτό. Εμείς κατά την χάραξη και εφαρμογή ε, πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπουμε σε συμβουλές από σημαντικούς παγκόσμιους φορείς όπως εσείς, όπως είπατε η αρμοστία του για τους πρόσφυγες για να διαμορφώσουμε την πολιτική μας. Όπως είπατε, ένα οργανωμένο και εύρυθμο πρόγραμμα επανεγκατάστασης δεν καταργεί τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο. Απλώς ε, παρέχει έναν τρόπο ε, για μια θετική εμπειρία, μια περίθαλψη των ε, ευάλωτων και αυτό χρειάζεται η Ευρώπη. Ε, μια θετική πλαισίωση χορήγησης προστασίας ε, στους χρήζοντες προστασία. Και όπως είπατε, η επανεγκατάσταση μας ανοίγει την πόρτα για να κάνουμε μια καλύτερη πλαισίωση αυτού του φαινομένου και ίσως θα μπορούσαμε να φανούμε και πιο ενωμένοι κατά τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου επανεγκατάστασης. Αμέσως μετά το θέμα αυτό θα εξετάσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πλαίσιο. Ε, είπατε όμως ότι θα πρέπει να γίνει εκ παραλλήλου συζήτηση για τη διαδικασία ένταξης και η ε, επανένταξη δίνει ευκαιρία για καλύτερο προγραμματισμό της ένταξης. Επίσης, τι γίνεται με τις αυθόρμητες αφήξεις και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να διδαχθούμε και να πρωτοστατήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση ε, αυτού του προβλήματος. Θα μπορούσατε να μας ε, δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις προτάσεις σας και επίσης ε, πώς λαμβάνετε υποθέσεις επανεγκατάστασης στις ΗΠΑ και ποιος είναι ο ρόλος, είπα, της αρμοστίας του ΙΕ για τα θέματα αυτά. Η κυρία Σοντόα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε κύριε Μίλιμπαντ για την πολύ ε, μεστή και ενημερωτική και διαφωτιστική παρουσίαση που μας κάνατε. Έχουμε χιλιάδες σελίδες ε, και χιλιάδες ώρες ενασχόληση με το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή που δυστυχώς πήγαν χαμένα όλα και έχουμε μεγάλες δυσκολίες ε, με το Συμβούλιο, γιατί όλα αυτά που επεξεργαστήκαμε και πολύ κοπιαστικά ε, εκπονήσαμε τους τελευταίους 20 και μήνες ε, πήγαν στο βρόντο εξαιτία της απροθυμίας του Συμβουλίου να τα εφαρμόσει. Επίσης, μιλάμε για άτομα που αντιμετωπίζουν ακραίες καταστάσεις, ιδιαίτερα ευάλωτα και χρήζουν προστασίας, διεθνούς βοήθειας και προστασίας. Και αυτό είναι ο ρόλος της ανάγκης προστασίας και της ασύλου. Αυτό το βλέπουμε και στα κέντρα καταγραφής, στα hot spots, που, όπου σειραίουν ασυνόδευτα παιδιά ανήλικοι που υπέστησαν το φοβερό τραύμα αυτής της δύσκολης μετάβασης και ε, έλευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει να αποφύγουμε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και να συνεχίσουμε μια συσσόρευση αυτών των τραυμάτων. Επίσης, από την επεξεργασία των υποθέσεων τον άσυλο στην Ιταλία και στην Ελλάδα, είδατε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και είπατε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε και στις χώρες προέλευσης. Αυτές οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις που εκδίδονται από τα προξενία, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο εύρυθμη διαδικασία για την εφαρμογή των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Η Σοράια πώς; Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μας πείτε συγκεκριμένα τι κάνετε ε, για το θέμα της ένταξης με τους πρόσφυγες στο Λίβανο, για παράδειγμα. Επίσης, Είχαμε και στα Βαλκάνια πολέμους και τα θύματα των πολέμων αυτών τα κυρίως οι Ρωμά που εστάλησαν στη Γερμανία, στην Ιταλία και ε, ενώ έχουν παραμείνει και 20 ετία ολόκληρη στη, στις χώρες αυτές εκδιώκονται και μένουν απάτριδες. Ασχολείστε καθόλου με το θέμα αυτό γιατί έχουμε παιδιά Ρωμά που έχουν γεννηθεί στην Γερμανία που έχουν μητρική γλώσσα τη γερμανική και εξαναγκάζονται να φύγουν να καταλήψουν τη χώρα με, απε, με αποπομπές απελάσεις. Επίσης στην Ιταλία έχουμε ενήλικες απάτριδες και άρα δεν έχουν δυνατότητα να λάβουν διαβατήριο ή να παρακολουθήσουν την επίσημη εκπαίδευση. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στιγμή γιατί μιλάμε για πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Η Σεσίλια Κέγκε. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις επί του θέματος. Έχουμε προσπαθήσει να σχεδιάσουμε προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάσταση, αλλά και για την επαναγκατάσταση. Ω τώρα δεν έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Όπως είδατε, του τελευταίους μήνες οι αφήξει έχουν ε, μάλιστα αυξηθεί στην Ιταλία. Οι αφήξει ε, ξεπερνούν τις προβλέψεις μας. Και ακόμα ε, την ευθύνη την έχουν οι χώρες πρώτης άφηξη. Βλέπουμε ο αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων να αυξάνεται εκρηκτικά. Όταν μιλάμε για τέτοια προγράμματα, είτε μιλάμε για μετεγκατάσταση, είτε για επαναγκατάσταση, πρέπει να έχουμε υπόψη και του ασυνόδευτου ανηλίκου. Ήθελα να ξέρω τι εγγυήσει δίδονται στι χώρε που παραλαμβάνουν αυτού του ανηλίκου και του υποδέχονται. Πώ εντάσσονται οι ανήλικοι στα προγράμματα αυτά και έπειτα για του ανθρωπιστικού διαδρόμου. Ποια είναι η δική σας ε, η συνεισφορά. Ο μόνος ανθρωπαστικός διάδρομος που έχει υλοποιηθεί έχει φτιαχτεί από την κοινωνία των πολιτών στην Ιταλία. Κάποιοι πολίτες ε, προχώρησαν σε ένα ανθρωπιστικό διάδρομο, έφτιαξαν ένα ανθρωπιστικό διάδρομο με μια έκθεση πρωτοβουλίας, ε, που τελικά με μια έκθεση πρωτοβουλίας τον εγκρίναμε εδώ εμείς στο κοινοβούλιο μας με ανθρωπιστικές θεωρήσεις αφού υποβλήθηκε το αίτημα. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να ενταχθεί στα προγράμματά σας, ώστε να υποφεληθούν και, αυτές, και άλλες χώρες από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Okay, thank you. And Mrs. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Κέγκε ε, ασχολείται, έχει την έκθεση για την ε, επαναγκατάσταση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και εσάς, David, για την παρουσία σας εδώ, θέλω να πω ότι η ε, κατάσταση είναι πολύ σημαντική για την ομάδα μου και για το κόμμα μου. Όμως δεν μπορούν να είναι αυτά δεσμευτικά για τις χώρες μέλη. Μόνο συστάσεις μπορούν να αποτελέσουν και προτροπές να υποδεχθούν πρόσφυγες. Αυτό ζητούμε εμείς και βλέπουμε ότι τουλάχιστον οι μισές χώρες μέλη δεν ανταποκρίνονται. Άρα σύσταση μεν ναι, επιβολή υποχρέωση όχι. Αλλά βεβαίω θεωρώ ότι οι χώρε πρέπει να λάβουν ευθύνε. Ντέβιντ, εσεί τοποθετηθήκατε. Είπατε ότι είναι κρίμα που αποχωρεί η Μεγάλη Βρετανία. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια σουηδική έξοδος. Ένα Brexit, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Τώρα, η ενδεχόμενη συνεργασία των χωρών του Περσικού κόλπου ε, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, που είναι οι πλουσιότερε χώρε του κόσμου. Δεν δέχονται όμω κανένα πρόσφυγα στο έδαφο του. Θα ήθελα να ακούσω κάτι σχετικό από εσά. Άλλο κανεί, λέει ο πρόεδρο. Γιάννα Γκόμε. Ευχαριστώ. Ερώτηση. Πώς κρίνεται την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. deal ας πούμε με την έννοια ότι δεν είναι συμφωνία είναι περισσότερο πώς να το πω κάπου τα βρήκανε εν τέλει επιστρέφονται στη Τουρκία άνθρωποι πριν καν να προλάβουν να καταθέσουν αιτήσεις ασύλου ποια είναι η γνώμη σας και για τη λίστα χωρών για αυτό το Ταμείο Trust μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας Λαβαλέτα Χαρτούμ με την Αιθιοπία πάνω πάνω στη λίστα. Η Αιθιοπία λαμβάνει πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκεί βοήθεια. Έχει όμως εκεί ένα καθεστώς το οποίο προβαίνει σε δολοφονίες ανθρώπων και προκαλεί έτσι κύματα προσφύγων και μεταναστών. Ποια είναι η αξιολόγηση που κάνετε. Ποτέ δεν θα ρωτήσω αν ε, υπάρχει άλλος κανείς ακόμη που θέλει, γιατί πάντοτε αυτό προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ, David. Ευχαριστώ ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. που θίγουν και ε, κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα και της νομοθετικής διαδικασίας. Θα προσπαθήσω να τις βάλω σε κάποια τάξη. Ερώτηση Κοέλιο. Μέχρι τώρα με έχουν κατηγορήσει για πολλά πράγματα, όχι για συντηρητικό. Το επίπεδο των 108.000 χρόνο, μήπως είναι υπερβολικά συγκρατημένο. Εγώ θεωρώ ρεαλιστικό να πάμε από τις 9.000 το χρόνο στις 108.000 το χρόνο σημαίνει μια σημαντική προσπάθεια στην πράξη. Δεν θα έλεγα ότι είναι το ελάχιστο το 108.000. Όμω, μια και τα Ενωμένα Έθνη μιλούν για 1.200.000 μέσα σε μια πενταετία, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεχτεί 500.000, κάτι τέτοιο μου φαίνεται είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα σπρώξει τι Ενωμένες Πολιτείες να κάνουν και αυτές κάτι για να έρθουν και αυτέ στο ίδιο ύψο. Δέχομαι ότι όντω είναι ρεαλιστική η πρόπτικη αυτή. Πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Και αν μπορώ να έρθω στην τελευταία ερώτηση τώρα για τον ρόλο των χωρών του Περσικού κόλπου. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν μηδέν υποδοχή προσφύγων, διότι οι χώρες αυτές δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης ή άλλες διεθνείς συνθήκες για την υποδοχή προσφύγων. Όμως υπάρχουν πολλοί Σύριοι, για παράδειγμα, Σαουδική Αραβία και στα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ρώτησα ποιο είναι το δικό μας επιχείρημα, ρωτήσατε μάλλον. Εγώ θεωρώ ότι οι χώρες αυτές πρέπει να υπογράψουν και μάλιστα επιγόντως τη Διεθνή Συνθήκη για τους πρόσφυγες και θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι οι Σύριοι που βρίσκονται στις χώρες αυτές, Σαουδική Αραβία και Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θεωρούνται μετανάστες, όχι πρόσφυγες, θα πρέπει οι χώρες αυτές όμως να δεχτούν και πρόσφυγες. Η σημασία, κατά τη γνώμη μας, της διατήρησης του ορισμού του πρόσφυγος και του συστήματος υποδοχής προσφύγων των πρωτοκόλων 1951 και 1962 που καθορίζουν το δικαίωμα, τα δικαιώματα μάλλον των προσφύγων Αυτά όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα δικαιώματα αυτά. Ένα τρόπος για να γίνει αυτό είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε κάποιον ο οποίος φεύγει από ένα τόπο για να σώσει τη ζωή του και έναν άλλο ο οποίος φεύγει για να βελτιώσει τη ζωή του. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός ο τελευταίος είναι κακός, αλλά είναι διαφορετικός, είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι σημαντικό επίσης και νομίζω ότι η έκθεση ΕΑΣΟ στην οποία αναφερθήκατε αναφέρεται σε αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα και οι αιτήσεις ασύλου, του, ασύλου τους. Έχουμε προσωπικό μας στην Ευρώπη, δεν περίμενα ποτέ να αναπτύξουμε προσωπικό στην Ευρώπη, έχουμε και ειδικέ προτάσεις για την ανάγκη ε, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους ε, νομομαθείς, περισσότερους διερμηνείς, περισσότερους ε, ανθρώπους για να μπορέσουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα. 50.000 αυτή τη στιγμή άνθρωποι που ζητούν άσυλο. Έχουμε πολλή εμπειρία. Ο ύπατος αρμοστής για τα, ΕΕ για τους πρόσφυγες κάνει τις σχετικές έρευνες και η καναδική κυβέρνηση που επιλέχθηκε την προηγούμενη χρονιά υποσχέθηκε να υποδεχθεί στην επικράτειά της 25.000 Σύρους πρόσφυγες. Το έπραξε αυτό μέσα σε 9 μήνες και με ομάδες τις οποίες επέλεξε ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών. Άρα το σύστημα υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Με ρωτήσατε αν έχουμε ιδιαίτερα προγράμματα για τους απάτριδες. Δεν έχουμε. Δεν έχω τίποτε ειδικότερα να σας πω εν προκειμένου. Σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, που ε, ρωτήσατε εσείς, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα από τα σκάνδαλα της περίοδου αυτής που διανύουμε. Θυμίζω και την περίπτωση του Καλέ. 900 παιδιά βρίσκονται εκεί, 500 ε, τα έχει δεχθεί καταρχήν το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν φτάσει όμως εκεί. Εγώ θεωρώ ότι οι υποθέσεις σαν αυτές είναι απαραίτητο να επιληθούν για να μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Το τελευταίο σχόλιο που είναι, αναφέρεται και στην πρώτη ερώτηση που ε, μου έθεσε η κυρία Σίπελ είναι η πολιτική απόχρωση. Αν ήμουν καλύτερο στα πολιτικά μπορεί να μην έκανα τούτη τη δουλειά που κάνω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά ο καλύτερος για να σας συμβουλεύσω για την πολιτική πτυχή ε, του θέματος. Τι να κάνετε δηλαδή για τα πολιτικά. Έχει σχέση αυτό και ε, με αυτό που ρώτησε η Μάρλιν Μπιόργκ. Το πλαίσιο δηλαδή μέσα στο οποίο κινείται η προσπάθεια αυτή. Εδώ μπορώ να σας πω δύο πρακτικά πράγματα. Αφενός δεν υπάρχει τίποτε το ισχυρότερο από τη μαρτυρία των ίδιων των προσφύγων. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και εσεί, ω εκλεγμένοι εκπρόσωποι και εγώ ω επικεφαλή μη κρατική οργάνωσης να δώσουμε φωνή στου πρόσφυγε. Είναι σαφέ πάντω, ότι οι πιο βαρύνουσε, οι πιο συναρπαστικέ, οι συναρπαστικές πιο έντονε ιστορίε, προέρχονται από τα ίδια τα άτομα εκείνα που διέφυγαν για να διασώσουν τη ζωή του. Δεύτερο, ένα θέμα το οποίο, ε, στο οποίο αναφέρθηκα χθε το βράδυ και προέρχεται από την Αμερικανική εμπειρία. 36 αμερικανικέ πολιτείε έχουν κυβερνήτες που δήλωσαν ότι δεν δέχονται στην επικράτειά τους σύρους. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο βέβαια. Οι πιο σημαντικές πολιτικές φωνές κατά των ανθρώπων αυτών προήλθαν από δημάρχους πόλεων που συχνά βρίσκονται σε πολιτείες που έχουν κυβερνήτες οι οποίοι λένε ότι δεν θα δεχθούν σύρους, όπως για το Τέξας για παράδειγμα, όπου οι δήμαρχοι του Χιούστον και Ντάλλας δήλωσαν ότι οι πόλεις τους θα παραμείνουν ανοιχτέ στους πρόσφυγες και στο μέλλον και στους ήρους επομένως. Και τέλος κάτι ακόμα, μια ευρύτερη, αν μου επιτρέπετε, σκέψη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσει μοναχά τα συμπτώματα της κρίσης του προσφυγικού, δεν πρόκειται να κερδίσει τις καρδιές και τα μυαλά των ψηφοφόρων. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην ρίζα του και βεβαίω και τα συμπτώματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η πηγή των διαφόρων συγκρούσεων είναι κατά περίπτωση διαφορετική, αλλιώτικη στο Αφγανιστάν, αλλιώτικη στη Σομαλία, στη Συρία και ούτω καθεξής. Αλλά θεωρώ ότι εκτός από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, η εμπλοκή με χώρες όπως Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία ε, είναι αναγκαία, όχι μόνο για να υπάρξει ε, μια απάντηση στο πλαίσιο της πολι... των πολιτικών που ασκούνται δηλαδή, αλλά και μια απάντηση πολιτική η απόφαση των Τούρκων να αντιμετωπίσουν τις ομάδες ε, λαθρεμπόρων είναι σημαντική και για του Τουρκούς και για τους Ευρωπαίους. Δεύτερο, βρισκόμαστε πληρώνουμε το τίμημα τώρα μια σειρά ετών όπου δεν συνομιλούσαν Ευρώπη και Τουρκία. Τρίτο, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό η μόνη λύση να είναι να ανταλλάσσονται πρόσφυγες από την Τουρκία με αυτούς και μάλιστα σε ε, ποσότητα ένα προς ένα που έχουν επιστραφεί. Στο κάτω της γραφής η Τουρκία τα τελευταία, δύο, ε, ε, ε, ε συγνώμη, τα πέντε χρόνια έχει υποδεχθεί 2,7 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες. Ίσως λέω με πολλά λόγια κάτι που θα μπορούσα να πω πιο σύντομα, δηλαδή ότι να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα στη ρίζα του και όχι μόνο τα συμπτώματά του είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ντέιβιτ. Ε, φαίνεται από τα χειροκρότηματα ε, πόσο εκτιμούμε και επικροτούμε το έργο σου. Ευχαριστώ τους βουλευτέ για τι ερωτήσει του και να σα πω ότι αμέσω μετά το δικό σου θέμα θα συζητήσουμε την πρόταση για το πλαίσιο επανακατάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω η, η συνεισφορά τη Διεθνού Επιτροπή Διάσωση μα έχει βοηθήσει πολύ. Η επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και η αποστολή τη αντιπροσωπεία στο Λίβανο και την Ιορδανία ε, είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης και θα συνεχιστεί η συνεργασία αυτή κατά την εκπόνηση της έκθεσης μας για την επανεγκατάσταση και την σχετική συζήτηση. Σε ευχαριστώ που μας αφιέρωσε το χρόνο σου και νομίζω ότι όλοι εκτιμήσαμε ιδιαίτερα σε αυτή την ευκαιρία που είχαμε για συζήτηση. Ευχαριστώ και πέραμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 4 της εμμερίσης διάταξης, το ενωσιακό πλαίσιο για την επανεγκατάσταση, παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά το, την παρουσίαση του πολύ αξιόλογου έργου της Διεθνούς Επιτροπής ε, Διάσωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας προτείνει την ε, τροποποίηση του κανονισμού 516-2014 για το νέο πλαίσιο επανεγκατάστασης ε, που συμπληρώνει το δεύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων του κοινού ευρωπαϊκού ασύλου και του σχετικού συστήματος. Και θέλουμε ένα εναρμονισμένο, διαρθρωμένο και μόνιμο πλαίσιο επανεγκατάσταση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ένα πρόγραμμα επανεγκατάσταση και δημοσίευσε σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ. Το 2015, μετά τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάσταση, το Συμβούλιο υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2015 τα συμπεράσματά του με απόφαση να επανεγκαταστήσει 22.000 και πρόσωπα ε, που χρήζουν ε, άμεσα προστασίας με βάση τις ε, οικειοθελείς υποσχέσεις των κρατών μελών. Με βάση την πέμπτη έκθεση επανεγκατάσταση, μόνο 8.000 άτομα έχουν επανεγκατασταθεί στα μέσα Ιουλίου. Άρα δεν είμαστε ούτε στα μέσα της υλοποίησης του στόχου. Ενώ ταυτόχρονα οι παγκόσμιε ανάγκε αυξάνονται και η δημιουργία ενό αποτελεσματικού συστήματο επανεγκατάσταση αποτελεί κεφαλαιόδη στόχο και μάλιστα είχαμε ήδη την ευκαιρία για προκαταρκτικές συζητήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα περιμένουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συζήτησης. Θα έχουμε το πρώτο πρόγραμμα επανεγκατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι άνευ προηγουμένου στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κύριε Νίλσεν, θα σας δώσω το λόγο και μετά θα ακούσουμε την εισηγήτρια και τους σκιώδης εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή την πρόταση που όπως είπατε θα καταστήσει την επανεγκατάσταση πιο ε, δομικό στοιχείο της ε, πολιτικής μας για το άσυλο και βασικό στοιχείο της πολιτικής αυτής ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους στόχους. Η πρόταση απαρτίζεται από τρεις στόχους. Καταρχήν, η παροχή νόμιμων και ασφαλών διάβλων προσφύγων χρηζών προστασία για να έρθουν στην Ένωση. Δεύτερον, συμβάλλει στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Και τρίτον, ε, επιτρέπει στην Ένωση να συμβάλλει σε διεθνείς σχετικές πρωτοβουλίες, ε, προσφέροντας ενιαίες υποσχέσεις ε, για την επανεγκατάσταση στα Ηνωμένα Έθνη. Τα βασικά συστατικά του πλαισίου είναι δύο Πρώτον, συμφωνία για ένα ετήσιο σχέδιο επανεγκατάστασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσδιορίσει τους συνολικούς αριθμούς προσφύγων ε, για επανεγκατάσταση το επόμενο έτος και η κατανομή ε, των αριθμών αυτών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τις βασικές γεωγραφικές προτεραιότητες, δηλαδή ε, σε ποιες περιφέρειες θα επικεντρωθούν τα σχέδια επανεγκατάστασης το πρόγραμμα επανεγκατάστασης ε, θα εφαρμοστεί μέσω ενός ή περισσότερων επιμέρους προγραμμάτων ε, ανάλογα με συγκεκριμένες χώρες, ε, περιοχές ή ομάδα πληθυσμού και θα προσδιορίζει με περισσότερες λεπτομέρειες την εφαρμογή της κατανομής στο συγκεκριμένο σχέδιο. Τώρα, για να δούμε πώς το πρόγραμμα και τα επιμέρους σχέδια θα εφαρμοστούν. Το πρώτο βήμα τη χρονιά πριν την θέσπιση αυτού του προγράμματος επανεγκατάστασης θα έχουμε διαβουλεύσεις που θα συγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ομάδα επανεγκατάστασης υψηλού επίπεδου με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, της ΕΕ των ΗΠΑ και την IOM. Αυτό θα κάνουμε του χρόνου για την επανεγκατάσταση. Καταρχήν θα δούμε ποιος θα είναι ο συνολικός στόχος για τους αριθμούς ε, των προσφύγων, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και πού θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας. Ανάλογα με τη συζήτηση στην ε, ε, Επιτροπή αυτή υψηλού επίπεδου θα προτείνουμε την υιοθέτηση μιας εφαρμοστικής απόφασης του Συμβουλίου που θα προσδιορίζει τους αριθμούς για το επόμενο έτος και τις γενικές γεωγραφικές προτεραιότητες. Εδώ τονίζουμε την ανάγκη για τη χρήση μιας απόφασης, εφαρμοστικής απόφασης του Συμβουλίου. Γιατί νομίζω ότι σε περίπτωση κατανομής των αριθμών καλύτερα να προσφύγουμε σε απόφαση του Συμβουλίου και όχι εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέτοια είδους απόφαση και θα καθορίζει το ετήσιο σχέδιο ε, το, της επανεγκατάστασης, αριθμούς και προτεραιότητες και ταυτόχρονα θα υποβάλλουμε και την πρόταση για τον ετήσιο προπολογισμό της Ένωσης με βάση την κανονική διαδικασία του προπολογισμού και στην πρόταση αυτή θα περιλαμβάνουμε και τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για να χρηματοδοθούν οι συγκεκριμένες επανακαταστάσεις που προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο του χρόνου αυτού. Η συμφωνία για το ίδιο το σχέδιο και για τον προπολογισμό του θα ε, δρομολογούνται εκ παραλίλου. Τέλος, προετοιμασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει ένα περισσότερο μία ή περισσότερες εφαρμοστικές αποφάσεις που θα προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα σχέδια επανεγκατάστασης που θα εφαρμόζουν αυτό το ενιαίο σχέδιο επανεγκατάστασης, μία ή περισσότερες εφαρμοστικές αποφάσεις θα εξαρτηθεί από το αν πρόκειται για συγκεκριμένη για μία μόνο χώρα και σίγουρα ε, θα δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες μας, αν έχουμε τρεις ε, περιοχές προτεραιότητες έχουμε τρία σχέδια επανεγκατάστασης, αλλά ε, θα είναι ελαστικό το πρόγραμμα ώστε να προσαρμοζόμαστε στις ετήσιες ανάγκες και συνθήκες. Για τον καθορισμό του προγράμματος αλλά και των επιμέρους σχεδίων επανεγκατάστασης ε, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά στοιχεία και παράγοντες. Για παράδειγμα, τον αριθμό των ατόμων που χρήζουν ε, διεθνούς προστασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα. Επίσης ε, διευρύνεται ο παραδοσιακός, ο τυπικός ορισμός της επανεγκατάστασης για να καλύψει και εσωτερικά εκτοπισμένους που χρήζουν διεθνούς προστασίες. δηλαδή όχι κατά ανάγκη ε, ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε άλλη χώρα, αλλά και εσωτερικά εκτοπισμένους. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους σχέδια θα αναζητήσουμε συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα διεθνούς επιχειρησιακής προστασίας στη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή και θα λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες επανεγκατάστασης και άλλων χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα εξετάσουμε και τις ε, γενικές μας σχέσεις συνεργασίας με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και τις προσπάθειες, η προθυμία της τρίτης χώρας να μειώσει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και την ε, επιθυμία να θεσπίσει το δικό του σύστημα ασύλου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες φυσικά θα ληφθούν υπόψη στο πρόγραμμα. Δεν σημαίνει ότι τέτοιου παράγοντε όπως η συνεργασία για τη μετανάστευση υποχρεωτικά θα αποτελούν τμήματα κάθε σχεδίου ή προγράμματος επανεγκατάστασης. Πιθανό να γίνει, θα εξεταστεί περιπτωσιολογικά και θα αποφασιστεί κάτι τέτοιο περιπτωσιολογικά. Τα δύο τελευταία στοιχεία. Τι προβλέπει η πρόταση. Προβλέπει μια σαφέστερη κοινή διαδικασία και κοινά κριτήρια για τη διαδικασία λήψη απόφασης επανεγκατάστασης. Τα αποφάσει δηλαδή που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για έναν υποψήφιο επανεγκατάσταση, το τι κριτήρια θα εφαρμόζουν, τι διαδικασία θα εφαρμόζουν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για το καθεστώς που θα δίνεται σε αυτό το άτομο, θα εμπίπτουν σε μια κοινή διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι άνευ προηγουμένου, γιατί δεν είχαμε μέχρι στιγμή τέτοιε κοινέ διαδικασίε και κοινά κριτήρια στην κοινοτική νομοθεσία. Βέβαια, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν είναι υπεύθυνα για τι μεμονωμένε αποφάσει. Προβλέπονται δύο είδη διαδικασιών. Τα σχέδια επανεγκατάσταση ε, προβλέπουν τι επιλογέ θα υιοθετηθούν σε κάθε σχέδιο. Έχουμε καταρχήν την κανονική ε, διαδικασία, την παραδοσιακή διαδικασία επανεγκατάσταση που εφαρμόζεται και σήμερα από τα κράτη-μέλη, που είναι κάπως πιο χρονοβόρα διαρκεί ένα με δύο χρόνια. Προτείνουμε σύνμιση αυτή τη διαδικασία, συντόμευση, αλλά είναι μια πιο διεξοδική για να καθοριστεί το καθεστώ που αποδίδεται στο συγκεκριμένο ετούντα και στη τελική ανάλυση για το καθεστώ πρόσφυγα. Η δεύτερη διαδικασία είναι η συνοπτική διαδικασία, είναι πιο γρήγορη επιταχυμένη διαδικασία. Εδώ εμπνεόμαστε από αυτό που κάνουν τώρα τα κράτη-μέλη σε σχέση με την Τουρκία και που ήταν αρκετά επιτυχημένο, γιατί οι αποφάσεις πλέον λαμβάνονται με το ταχύτερο και συνοπτικότερο τρόπο. Έχουμε λοιπόν διαδικασίες, την κλασική, την κανονική και την συνοπτική, την ταχύτερη. Και επίσης ε, ε, με την συνοπτική διαδικασία δίνει το καθεστώς ε, προστα... παροχής προστασίας, όχι πρόσφυγα. Θα εξαρτηθεί από το, στόχο για το τι, τι διαδικασία θα εφαρμοστεί. Πάντως γίνεται εναρμονισμένη η εφαρμογή των διαδικασιών. Προτείνουμε επίσης 10.000 ε, ευρώ εφάπαξ ποσό για κάθε άτομο που θα έχει υποφεληθεί από την επανεκατάσταση και επίσης ε, προτείνουμε και κάποιες τεχνικές αλλαγές στον κανονισμό για τα κονδύλια του ΑΜΙΦ, οπότε να προσαρμοστούν τα κονδύλια αυτά στο νέο σύστημα και πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και την κατανομή των οικονομικών πόρων για κάθε σχέδιο επανεγκατάστασης, αυτό θα ακολουθήσει τη συνήθη δημοσιονομική διαδικασία και θα γίνει παράλληλα με τον καθορισμό του ετήσιου προγράμματος επανεγκατάστασης και των επιμέρους σχεδίων επανεγκατάστασης. Αυτά ως προς τις αδρές γραμμές του, της πρότασης και περιμένω τις ερωτήσεις Ευχαριστώ. Θα έρθω αμέσω στον εισηγητή. Βλέπω και παρουσία σκιωδών εισηγητών. Την εισηγήτρια εννοώ βέβαια. Μαρλίν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω λέγοντας ότι υπήρξε προτεραιότητα για το Ευρωκοινοβούλιο η εξέβρεση νόμιμων τρόπων για να ε, φτάσουν εδώ οι, ε, οι ε, πρόσφυγες. Η μετεγκατάσταση είναι ο πιο καλά θεμελιωμένος τρόπος. Έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο το διαχειρίζεται ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών και οι συμμετέχοντες έχουν δείξει βεβαίως και έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και για την ένταξη. Χώρες όπως οι Ενωμένες Πολιτείε υποδέχονται 85.000 τον χρόνο. Και αυτό είναι προφανές ότι και, είναι προφανές εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει την προσπάθεια. Έχει λοιπόν προστιθέμενη αξία το πρόγραμμα πρέπει όμως να δείξουμε, πρέπει όμως να επιτύχουμε σημαντική αύξηση των αριθμών. Να δείξουμε αλληλεγγύη σε μια δύσκολη κατάσταση και επίσης να ε, αυξήσουμε την ποιότητα. Πολλές χώρες μελή έχουν καλές εμπειρίες και καλή ιστορία σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρώπη να βασιστεί σε αυτές τις εμπειρίες και να βελτιώσει την υποδοχή. Εν ώψη του ιστορικού αυτού, είναι σαφές ότι χρειάζεται ενίσχυση οι προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας τις αρχές και την ιστορία επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων μετεγκατάστασης, εγώ έχω κάποιες ανησυχίες σχετικά με την πρόταση που γίνεται. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τονίσω ορισμένες από τις πιο βασικές ανησυχίες και να ζητήσω και κάποιες διευκρινήσεις. Το πρώτο και προφανές είναι ότι στην πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γράφει ότι πρόκειται για μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στο άρθρο 4 λέει ότι τρίτε, η, η, η, πραγματική συνεργασία για τη διαχείριση των συνόρων τρίτων χωρών είναι σημαντικό. Στην ουσία δηλαδή φέρνουν τη συμφωνία με την Τουρκία να την κάνουν νόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικρίνει τη συμφωνία με την Τουρκία. Δεν είναι ο σωστό τρόπο ούτε για τη μετεκατάσταση ούτε για ε, να κινηθούμε προ τα εμπρό. Χρειάζεται ένα διαφορετικό πλαίσιο με συνεργασία και το Συμβούλιο. Και αυτά τα τόνισε και ο Μίλιμπαντ προηγουμένω, αλλά και άλλοι με του οποίου έχω συνομιλήσει, ότι εδώ ε, το πλαίσιο αυτό είναι προβληματικό. Άλλο πρόβλημα είναι η επανένωση οικογενειών. Υπάρχει σχετική νομοθεσία όμως της Ένωσης για τον τομέα αυτό, εφόσον το έχουμε. Και αν ε, μείνουμε στις 20.000, για τη μετεκατάσταση. δεν θα υπάρχουν καν αρκετοί για να γίνει και η οικογενειακή επανένωση. Δεν είναι λοιπόν ε, αποδεκτή αυτή η λύση. Πρέπει να ζητήσουμε οι χώρες μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Κριτήρια τώρα. Άνθρωποι που είναι ευάλωτοι κοινωνικο-οικονομικά Νομίζω ότι όντως χρειάζεται μια ευρύτερη θεώρηση των ομάδων, όμως η έκθεση αναφέρεται περισσότερο σε έλεγχο και λιγότερο σε προστασία. Σας ερωτώ, τι εννοειται οταν όταν λέτε ε, κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτα τα άτομα. Άλλο πρόβλημα είναι οι λόγοι αποκλεισμού. Η πρόταση αυτή τιμωρεί εντό εισαγωγικών του ανθρώπου οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν και εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιμωρούνται αυτοί δεν θα τους επιτρέπουν δηλαδή να συμμετέχουν σε προγράμματα μετεγκατάστασης για μια πενταετία. Αυτή η κατασταλτική διάθεση μου φαίνεται δεν είναι σωστή. Εάν μια χώρα μέλος απορρίψει έναν που ε, πηγαίνει για μετεγκατάσταση, τότε τον απορρίπτουν όλες οι χώρες μέλη ενώ οι χώρες μέλη μπορεί να έχουν διαφορετική, ε, διαφορετικούς λόγους όπως ε, δεν μπορούν για παράδειγμα να προσφέρουν ε, την απαραίτητη φροντίδα υγείας. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι ρόλοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όμως, ανησυχώ ότι ο ύπατος αρμοστής των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες θα πρέπει να διατηρήσει ισχυρό ρόλο και αυτό δεν συμβαίνει εδώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν, μπορεί να, δεν είναι σωστό να υπάρξει ε, επικάλυψη ε, των ε, δομών, δηλαδή να δημιουργήσουμε και εμείς παράλληλε δομές με τον ύπατο αρμοστή. Θέλω να ρωτήσω επίσης με ποιον τρόπο το πρόγραμμα θα συμπληρώσει αντί να κινείται παράλληλα με τεχνικά προγράμματα. Λέτε στο προήμιο, στο 31, ότι δεν επηρεάζονται τα εθνικά προγράμματα των χωρών μελών. Εγώ όμω πιστεύω ότι αυτό θα γίνει, δηλαδή θα επηρεαστούν. Και ο φόβος είναι ότι οι φυστάμενα εθνικά προγράμματα απλά θα ενταχθούν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και τελικώς θα μειωθούν αντί να αυξηθούν οι αριθμοί των ατόμων, ατόμων που μετεγκαθίστανται. Ευχαριστώ να ακούσω και από τους κοιόδη ηγητές τι απόψει του να μην λησμονούμε όμω ότι πρέπει τελικώ να αυξηθεί ο αριθμό των μετεγκαθισταμένων και η ποιότητα τη μετεγκατάστασης. Αυτό πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό, διότι το πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε. Πρέπει να δείξουμε ότι με τον τρόπο αυτό φροντίζουμε για τι ανάγκε των ανθρώπων αυτών. Και ο διορθώνει, μιλούμε για επανεγκατάσταση και όχι για μετεγκατάσταση. Εγώ θα περιλάβω στη διαδικασία όλους τους βασικούς παράγοντε, βασικούς παίκτε, βεβαίω και το Συμβούλιο, αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνεργαστώ με του κοιόδης εισηγητές και εισηγητρίες για να ε, συντάξουμε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάλιν. Να περάσουμε ευθύ αμέσω στου κύριου συζητητέ. Ο κύριο Ντία μέρα δεν μπορούσε να είναι εδώ για το ΕΛΚ. Οπότε λόγο στην κυρία Πύρη για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε. Νομίζω ότι η επανεκατάσταση είναι η μια απόκριση για την ε, κρίση των προσφύγων με έναν τρόπο αξιοπρεπή. Παρά τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τον αριθμό των τον άσυλο πέρσι, ο αριθμό των ανθρώπων που έχουμε επανεγκαταστήσει είναι πραγματικά ένα αριθμό τελείω ανεπαρκή που μα ντροπιάζει. Όπω είπε κάποιο, είναι ένα παράδειγμα η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, όπου η επανεγκατάσταση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, όμω ένα εξάμεινο έχουμε δώσει σε χίλιους πρόσφυγες μόνο με ασφαλή πρόσβαση. Εδώ λοιπόν, επί της αρχής, χαίρομαι πολύ που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν κανονισμό περί επανεγκατάσταση. όμω το ερώτημα είναι εάν πρόκειται να αυξηθεί ο ρυθμό επανεγκαταστάσεων των πλέον ευάλωτων προσφύγων προ την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτή είναι η καθοριστική ερώτηση. Διότι αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε ποιο ο λόγος της πρότασης αυτή καθεαυτής. Ναι, και για στοιχεία που δεν αναφέρει η πρόταση. Κατάλαβα καλά ότι εάν από τα προγράμματα του EMIF δεν αυξηθεί ο προπολογισμός και για κάθε επανεγκαθιστούμενο παίρνει μια χώρα 1000 ευρώ, παρόλα αυτά παραμένει ένα πλαφόν στην πρόταση, μια, ένα νοτατόριο. Ποιο είναι αυτό το νοτατόριο λοιπόν ή χρειάζεται νέος κανονισμός ή απλώς ένας μεγαλύτερος προπολογισμό και να πιέσουμε τα κρατη να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο επανεγκατάστασης. Μια άλλη ερώτηση είναι η εξής. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιε είναι οι παγιωμένε πρακτικέ για την υλοποίηση του προγράμματο επαναγκατάσταση και βάσει τη δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Έχω υποβάλει γραπτή ερώτηση προ τον Επιτροπό Αβραμόπουλο και λέγεται ότι δεν μπορούν ε, να κοινοποιηθούν αυτέ οι παγιωμένε πρακτικέ στο Κοινοβούλιο, αλλά εφόσον μα υποβάλλεται μια τέτοια πρόταση, ε, το βρίσκω λίγο προφανέ. Αυτέ οι πρακτικέ μάλλον πρέπει να γνωστοποιηθούν και στο Κοινοβούλιο, αν θέλουμε να είμαστε προσεκτική στην εξέταση και υπεύθυνη στην εξέταση του κανονισμού. Έπειτα πώ θα εμπλέξουμε στην όλη διαδικασία με ενεργό τρόπο την κοινωνία των πολιτών. Ε, δεν βλέπω κάτι σχετικό στην πρόταση αυτή τη στιγμή. Και μετά ακόμη ένα ζωτικό ερώτημα. Γιατί να διασυνδέσουμε την επανεγκατάσταση ευάλωτων προσφύγων με το κατά πόσον οι χώρες υποδοχής ε, αντιμετωπίζουν τις παράνομες ε, μεταβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χρησιμοποιεί ένα ανθρωπιστικό εργαλείο, σαραβδί, για να χτυπήσουμε την ευρωπαϊκή Νομίζω ότι το ευάλωτο των προσφύγων δεν μπορεί να σχετιστεί με τον έλεγχο των σύνορων από τι χώρε υποδοχή. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει λίγα περισσότερα. Αυτή η πρόταση, κατά την άποψή σα, είναι ανθρώπινη. Ε, έχει σκοπό να αυξήσει όντω τον αριθμό των επανεγκαταστάσεων προ την Ευρώπη. Ιδάλλως, για να είμαι τελείω ειλικρινή, δεν βλέπω και μεγάλη ανάγκη για αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κέιτι οι υπόλοιποι συγκητές που είναι εδώ για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Ντεπρέ. Ζεράλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι η εισηγητής ε, εγώ ίδιος, ο κύριος Μισελ είναι ο υπεύθυνο, αλλά με παρακάλεσε να σας διαβιβάσω τις σημειώσεις του. Να σας τη διαβάσω δηλαδή. Αγαπητά, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μπιόρκ. Ο κύριος Μισελ ανυπομονεί ε, να συνεργαστεί μαζί της και με τους υπόλοιπους κοιόδης εισηγητές. Χαιρόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους προβλέπει ένα νόμιμο πλαίσιο για τη μετανάστευση και η πρόταση αυτή προτείνει εφ' εξής μία ε, επίσημη εναλλεκτική για να μην υπάρχουν επικίνδυνα και θανατηφόρα ταξίδια προς την Ευρώπη. Ο μηχανισμό αυτό πρέπει να γίνει μια από τι σοβαρότερε αποκρίσει στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που συχνά είναι χαοτική και να δώσει αξιόπιστε εναλλακτικέ στα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονται τι ανθρώπινε ζωέ. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει τα ωριά τη. Κάποια στοιχεία δεν ε, ε, δείχνουν ότι θα λειτουργήσει με τρόπο αποτελεσματικό ο μηχανισμό αυτό. Οι λεπτομέρειε τη πρόταση δεν θα θίξω, θα κάνω απλώ τρει διαπιστώσει. Πρώτον, ε, πραγματικά ευνηδιάζομαι από τον ελάχιστο, για να μην περιφερειακό ρόλο, που θα διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Μετανάστευση. Ε, μια ευρωπαϊκή διάσταση κρίση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει δυναμική κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού ε, Οργανισμού και θα έπρεπε να αναλάβει ως φορέας κλειδί στην όλη διαδικασία. Δύο. Επιπλέον, ε, αφού το Συμβούλιο αποφάσισε μόνο του ποιε θα είναι οι δεσμεύσει που θα λάβει το κάθε κράτο μέλο χωρί την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου, αναρωτιέμαι πού βρίσκεται το θεμητό και το ένομο τη ε, πολιτική αυτή. Και τρίτον, πιστεύω ότι οι 10.000 ευρώ που προβλέπονται από το Ταμείο δεν είναι επαρκέ κίνητρο για τα κράτη-μέλη ώστε να γίνει ο μηχανισμό αυτό μια βιώσιμη λύση. Ακόμη περισσότερο, διότι βρισκόμαστε καθυλωμένοι από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που περιορίζεται από το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ανώτατο όριο θα πρέπει να προβλεφθεί για την επανεγκατάσταση από το σχετικό ταμείο και προβλέπει για τις τωρινές δημοσιονομικές πρόπτικες 300, 300 εκατομμύρια ευρώ στο 2020. Δηλαδή περίπου 36.000 άτομα που θα μπορούν να επανεγκατασταθούν. Και ε, σημειώνω ότι επιπλέον ο κύριος Μισελ ε, προτείνει να είμαστε πιο αισιόδοξοι και να αναζητήσουμε απαντήσεις που θα είναι πολύ σημαντικές για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος. Τώρα και εγώ να θέσω δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτη, όπως το θύμισα, το ανώτατο όριο του χαρτοφυλακίου του ε, Ταμείου για το άσυλο και τους μετανάστες καθώς και την ενταξή τους, το ΑΜΙΦ τι όρια προβλέπετε για το μέλλον, εφόσον θα υπάρξει ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων επανεγκατάστασης. Και μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε, είδα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είδα ότι θα φορολογηθούν τα κράτη που θα αρνηθούν ε, την ποσόστοση προσφύγων που τους αναλογεί βάσει του μηχανισμού της Επιτροπής. Είναι λογικό αυτό. δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, εάν ε, χρησιμοποιήσαμε αυτά τα ποσά για να χρηματοδοτήσουμε το ταμείο αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Προβλέπεται ότι το Συμβούλιο θα πρέπει ετησίω να συμφωνεί ω προ την ποσόστοση των, του αριθμού των ανθρώπων που θα επαναγκαθίσταται ε, και αυτό με, την, με μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτό προτείνει ο κανονισμό. Η συνθήκη προτείνει στο άρθρο 221 όμω ότι αυτό είναι αποκλειστική, αρμο, ε, ότι αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ε, της Επιτροπής. Ε, εδώ πρέπει να δούμε ε, τι είναι η ε, αρμοδιότητα του Συμβουλίου, αν είναι κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα ή όχι. Εγώ καλά τα έχω καταλάβει. Θα πρέπει να υπάρχει εκτελεστική πράξη ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε αλλά οι, ερωτη... απαντήσεις θα δοθούν στο τέλος. Ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Μισελ για το μήνυμα στην αρχή. Στη συνέχεια. Για τους Πρασίνους, η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαια ότι μιλούμε για ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης ή ένα νέο ε, νομοθέτημα για να περιορίσουμε και πάλι την εισρωή προσφύγων ε, στην Ευρώπη και να βάλουμε κάποιους όρους, γιατί επιτάπητος έχουμε μία πρόταση που δεν λαμβάνει υπόψη τον ορισμό της Γενέβης για τους ε, πρόσφυγες, αλλά ε, περιλαμβάνει και την οικογενειακή επανένωση ακόμη και Ευρωπαίων υπηκοών και των συζύγων τους. Δηλαδή, αν θέλω να φέρω έναν αλλά ε, πω σύντροφο θα θεωρηθεί σε επανένωση. Επίσης, τα 10.000 ευρώ ανά πρόσωπο. Δεν ξέρω ότι αυτό συνάδουμε την αρχή της επανεγκατάστασης. Θα έχουμε και κοινωνικο-οικονομικά θέματα. δεν νομίζω όμως μια τέτοια πρόταση να περάσει αυτό στο κοινό και που δεν ξέρει τι εστί πολιτικός ε, πρόσφυγας. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιους όρους τρίτες χώρες με πρόσφυγες που είναι επιλέξιμοι για επανεγκατάσταση στις χώρες αυτές μπορούν να υποφεληθούν από την επανεγκατάσταση στην Ευρώπη μόνο αν συμφωνούν με, την, με τις αρχές της συμφωνίας της επανεισδοχής. Επίσης, μιλήστε για εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δηλαδή θα αποφασίζει κάθε χρόνο τι περιοχές θα είναι επιλέξιμες για επανεγκατάσταση και θα το χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής. Αυτά όμως δεν είναι ελάχιστες προϋποθέσεις επανεγκατάστασης, αλλά μέγιστες. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα καταφέρουν να συμφωνήσουν για τέτοιου είδους αρχές. Γιατί πρόκειται για ένα ανώτατο όριο που θα τους δεσμεύσει, που είναι ο προϋπολογισμός. Εγώ προτιμώ να επικεντρωθούμε στα ελάχιστα και μόνο 14 χώρες έχουν μέχρι στιγμής προγράμματα επανεγκατάστασης, άλλες 14 δεν έχουν. Επίσης, πού είναι η ε, μελέτη επιπτώσεων και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 14 ε, χώρες που δεν έχουν προγράμματα επανεγκατάστασης. Μήπως έτσι υποβαθμίζουμε, υποβιβάζουμε τις προδιαγραφές επανεγκατάστασης για τις χώρες που ήδη εφαρμόζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι οδυνηρό να πλησιάζουμε προς τη μεγάλη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής ε, κρίσης και να αναζητούμε ακόμη υποσχέσεις ε, για επανεγκατάσταση ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει ακόμη τις προσφορές, δεν έχει κάνει υποσχέσεις περισσότερο επικεντρώνεται στις επιστροφές. Νομίζω ότι είναι δύσκολο και πολύ προβληματικό να μετατρέψουν αυτή την πρόταση επαναγκατάσταση πραγματικά ανθρωπιστική πρόταση. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει η συγκήτρια, πάντως δεν προσβλέπουμε αδημονία στον τριμερή διάλογο. Ο κύριος Κοράου, που είναι και συγκητής του EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινάω από την προπόθεση ότι συμφωνούμε με την ιδέα να υπάρχει ένα πρόγραμμα επαναγκατάσταση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται ένα ανθρωπαστικό εργαλείο για νόμιμη πρόσβαση στη διεθνή προστασία και αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Βεβαίω, η πρόβλεψη στήριξη 10.000 ευρώ ανά άτομο που επαναγκαθίσταται είναι ένα κίνητρο για τα κατημέλη και ελπίζουμε να αυξηθεί ο αριθμό των επαναγκαθιστούμενων ε, ώστε να αγκαλιάσουν το πρόγραμμα αυτό και τα κάτι μέλη που τώρα έχουν αρνηθεί να παρακαταστήσουν στο έδαφο του πρόσφυγε. Όμω, με ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο που τόσο πολύ δεν έχει δώσει αποτελέσματα ω τώρα, ε, αμφιβάλλουμε για το πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλλει ένα τέτοιο πρόγραμμα και να το εφαρμόσει φαίνεται να είναι ένα εργαλείο διαχείριση τη μετανάστευση και όχι ένα εργαλείο πραγματικά ανθρωπιστικό, έτσι όπω προτείνεται. Δεν έχουμε αμφιβολίε για την προστιθέμενη αξία του προγράμματο σε σχέση με την τωρινή μορφή, όμω φοβούμαστε ότι μπορεί να πετύχει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να υποβαθμιστούν τα πρότυπα που υπάρχουν έτσι και αλλιώ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αύξηση στον αριθμό των αντόμων που θα επανακαθιστούν ίσα ίσα που ε, προβλέπεται ένας ελάχιστος αριθμό όπω όπως ε, επιβάλλεται από τι πιέσει του προπολογισμού και ένας ελάχιστος αριθμός ε, εφαρμόζεται με την οικογενειακή επανένωση αλλά το Συμβούλιο χρησιμοποιεί το μηχανισμό της επικουρικής στήριξης και βεβαίως δεν θα μειωθεί ο ρυθμός αυτών που πέφτουν στη θάλασσα για να ταξιδέψουν μέσα στην απελπισία τους. Με την επανεγκατάσταση επίσης, τα κράτη που έχουν δείξει την διάθεση συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προστατεύουν τα σύνορά τους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να προστατεύονται τα σύνορα αυτών που ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Ε, η κριτική μεταχείριση κατά ορισμένων κατηγοριών προσφύγων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι από χώρε προτεραιότητα δεν θα λαμβάνεται επαρκώ υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα οι υπόλοιποι συνάδελφοι για σύντομα σχόλια. Κυρία Γκόμνας. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις ανησυχίες των διαφόρων συναδέλφων και της ίδρυας σχετικά με το πώς και για πόσο καιρό ο ανθρωπιστικός σκοπός θα συνδέει την επανεγκατάσταση με τον, με την, με την, με τον των συνόρων από τρίτες χώρες και είναι και το παράδειγμα του Trust Fund που καταβάλει χρήματα σε ένα τρομερό καθεστώς το οποίο με τη σειρά του προκαλεί ρεύματα προσφύγων και μεταναστών και μιλώ για την Αιθιοπία της οποίας το αιθιοπικό καθεστώς το οποίο καθεστώς ε, σκοτώνει ανθρώπους επίσης βλέπω όπως ελέγχθηκε από την εισηγήτρια ότι πρόκειται για μια προσπάθεια κωδικοποίησης αυτής της, αδιαφανής, της αδιαφανούς συγγνώμη, συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ενώσης Τουρκίας. Διερωτώ με γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταυτού δεν εξετάζει τον τρόπο και διδάσκεται τα διδάγματα από τον τρόπο που δεν λειτουργεί η διαδικασία επανεγκαταστάσεως όπως θα έπρεπε και βεβαίω όχι μόνο για πρόσωπα που έρχονται από τρίτες χώρες και έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μεταξύ χώρων μελών της Ένωσης παρά τι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και παρά το γεγονό ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας επίγουσα καταστάσεω. και δεν μιλώ για νέε ε, χώρες μελιό που μία από αυτές δεν δέχονται ε, δεν δέχεται, ε, να, δεν πρόσφυγες μιλώ για τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Πορτογαλίας που δεν λειτουργεί. ανθρώπου από την ε, κοινότητα των Γεσίδη που έγιναν δεκτοί στην Πορτογαλία και παρόλα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα δεν έρχονται. Γιατί δεν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Η Πορτογαλία είπε κάτι επανάληψη είναι ότι είναι διατεθειμένη να υποδεχθεί του ανθρώπου αυτού. Και γνωρίζουμε οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται, ποιοι είναι κτλ. Επίση δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν εγκύπτει και στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων που γνωρίζουμε τόσοι πολλοί αγνοούνται ε, εν τω μεταξύ. Δεν λειτουργεί καθόλου επίσης η επανένωση οικογενειών. Οι χώρες μέλη επιλέγουν. Έλαβα μάλιστα πρόσφατα πληροφορίες ότι η Ιρλανδία ζήτησε να υποδεχτεί 10 χριστιανικές οικογένειες από την Συρία, να τις ε, φέρει δηλαδή στο ελληνικό έδαφος από την Ελλάδα. Ε, ε, πρέπει να βγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, διότι είναι αντίθετα και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και αντίθετα με τις ηθικές μας υποχρώσεις. Εν τέλει, θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι η προστιθέμενη αξία του κειμένου σας. που υποτίθεται ότι ε, βελτιώνει, αποκαθιστά ε, νόμιμους διάβλους για την έλευση των ανθρώπων. Ε, είναι όλα στα χέρια του, είπα, το αρμοστή των Ενωμένων για τους πρόσφυγες. Έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην καταλήγουν στα χέρια των λαθροδιακινητών. Η Μάριο. Ευχαριστώ. και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσίαση. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, ε, τις ψηφιακές τεχνολογίες για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες καταγραφής, ένταξης, πρόσβασης στην αγορά εργασίας να συντομεύσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Ξέρω ότι η Σουηδία και άλλες χώρες εφαρμόζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Γιατί δεν το γενικεύουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην επεξεργασία των αιτήσεων. Επίσης το μείζον ζήτημα είναι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πώς εξασφαλίσει το νέο σχέδιο επανεγκατάστασης στην πρόσβαση και στην αγορά εργασίας. Το είπαμε και τις προάλλες. Με τα επιμέρους σχέδια θα δημιουργηθούν κάποιες καταστάσεις που οι εργοδότες ε, δεν θα ενδιαφέρονται να προσλάβουν μόνο βραχυπρόθεσμα για βραχυπρόθεσμες ε, συμβάσεις εργαζομένους. Επίσης, κατάρτιση επαγγελματική θα προβλεφθεί. Και τι γίνεται με το κονδύλιο των 10.000 αναπρόσωπο. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χρήματα αυτά. Πώς θα εξασφαλίζεται ο έλεγχος, γιατί το βασικό έργο το επιτελούν ε, οι δήμοι, οι κοινότητες. Θα μπορέσουν αυτές να διαχειριστούν άμεσα τα κονδύλια ή θα πρέπει να περνάνε από την κυβέρνηση, από την κεντρική διοίκηση. Τι γίνεται με την πρόσβαση στην παιδεία, παιδεία κοινωνικό έργο είναι αρμοδιότητες των Δήμων. Γιατί να μην έχουν αυτές, αυτή η άμεση διαχείριση των κονδυλίων. Επίσης, ε, τι γίνεται με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Παρόλο που αυτές περισσότερο αναμειγνύονται και δραστηριοποιούνται, ε, συμμετέχουν ελάχιστα στις διαβουλεύσεις. Δεν θα μπορούσαν και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, να χρησιμοποιήσουν, να διαχειρίζονται τέτοια κονδύλια. Σας ευχαριστώ κυρία Γουνμπερκ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Η ιδέα είναι καλή. Και είπα ότι θα μπορούσαμε να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να υποδεχθούν, να περιθάψουν πρόσφυγες και να τους βοηθήσουν. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη με ένα δεσμευτικό μηχανισμό να χορηγήσουν προστασία. Όπως είπε η Μάλιν Μπιόρκ, το θέμα των κριτηρίων είναι ε, προβληματικό. Ε, οικονομική, κοινωνικο-οικονομική ευπάθεια, τι ακριβώς εννοείται. Επίσης, ε, οι συνθήκες, ε, το πλαίσιο που επηρεάζουν τη λήψη απόφασης. Πώς όμως θα ξεκαθαρίσουμε τι συνθήκε επικρατούν και στι 28 χώρε μέλη. Και τι γίνεται με τις ε, χώρε που δεν τηρούν καν τα κριτήρια της Κοπεχάγη. Δεν ξέρω πόσες φορές άκουσα την Άννα Γκόμες να μιλάει για τις ανοιχτές αγκάλες της Πορτογαλίας προς τους πρόσφυγες. Να σας στείλουμε 50.000 Πρόσφυγε από τη Σουηδία στην Πορτογαλία. Πολύ ευχαρίστω να του θέλετε. Γιατί δεν το κάνουμε όμω αφού είστε τόσο πρόθυμοι. Ο πρόεδρο. Και επανέρχομαι τώρα στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρόλο που πιέζει ο χρόνο, ακούστηκαν πολύ σημαντικέ ερωτήσει και από τους ηγητέ και από του ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα λοιπόν να σα δώσω όσο χρόνο χρειάζεται για να απαντήσετε τουλάχιστον στα βασικά ερωτήματα τι εισηγήτριας και ίσω και των σκιωδών. Παρακαλώ. Έχετε όσο χρόνο θέλετε. Σα ευχαριστώ. Ε, ας ξεκινήσουμε με τους αριθμούς των προσφύγων. Είναι... Ε, εννοείται ότι φυσικά θέλουμε να αυξήσουμε, είναι αυτονόητο θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των προσώπων που θα επανακαταστήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανεπαρκής ο αριθμός μέχρι στιγμής. Είπατε ότι δεν μπορούμε νομοθετικά να επιβάλλουμε ε, υψηλότερους αριθμούς και όντως σε αυτό το στάδιο δεν έχει οριμάσει η κατάσταση για κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να αποφασίζουν και περιπτωσιολογικά να κρίνουν πόσους θα δέχονται. Γι' αυτό και δεν έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς στην πρόταση. Πάντω πιστεύω ότι με το σχέδιο επανακατάσταση, το πρόγραμμα επανακατάστασης θα υλοποιήσουμε το στόχο και τη αύξηση του αριθμού. Καταρχήν να δούμε τι έχουμε σήμερα. Τίποτα δεν έχουμε σήμερα, γιατί είπατε να συγκρίνουμε με την παρούσα κατάσταση. Δεν έχουμε τίποτα, τίποτα που να, να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν, έσω, να συζητήσουν το θέμα της επανεγκατάστασης. Επαφείται στη διακριτική του ευχαίρεια και στην καλή του θέληση αν θέλουν να το κάνουν φέτος ή του χρόνου. Αν δεν θέλουν όμως δεν είναι υποχρεωμένοι. Ενώ τώρα τουλάχιστον έχουμε ένα πλαίσιο που προβλέπει δέσμευση των κρατών μελών και, τις κράτες ε, και των κρατών μελών κάθε χρόνο να θεσπίζεται ετήσιο πρόγραμμα επανεγκατάστασης, άσχετα αν περιλαμβάνει υψηλούς ή χαμηλότερους αριθμούς. Θα το αποφασίζουν αυτό τα κράτη-μέλη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πυροδοτήσει τη διαδικασία. Εμείς θα ξεκινήσουμε τις ε, συζητήσει στην Επιτροπή Ψηλού Επιπέδου και την πρόταση στο Συμβούλιο να καθορίσει αριθμού. Οπότε κάθε χρόνο το Συμβούλιο θα βλέπει αυτό το θέμα ε, στην ημερήσια διάταξη, δεν μπορεί να εθελοτυφλεί να κάνει πως δεν υπάρχει. Βέβαια δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα αυξηθούν οι αριθμοί των προσφύγων προς επανεγκατάσταση ή πώς θα καταφέρουμε να τους αυξήσουμε. Επίσης, ένα συναφές θέμα, το θέμα της διαδικασίας. Κύριε Ντεπρέ, έχετε δίκιο όπω συνήθω. Πάντως, εδώ έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες και ε, ε, δικαιολογείται η προσφυγή στην έκτακτη διαδικασία της εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου αυτή τη φορά. Γιατί επειδή η επανεκατάσταση γίνει στην, στην επικράτεια ενός κράτους, δικαιολογείται η ε, εξαίρεση για εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου. Για τον προϋπολογισμό πολλές ερωτήσεις και σχόλια, πάντως ε, γενικώ έχετε δίκιο ότι σίγουρα ανάλογα με τα κονδύλια που έχουμε θα δούμε και το εύρος του προγράμματος επανεγκατάστασης. Τώρα προτείνουμε 10.000 αναπρόσωπο και ισχύει εδώ το ίδιο ποσό και η διαρχή. Αλλά από εσά εξαρτάται από την αρμόδια για το δημοσιονομικό προπολογισμό αρχή να κρίνετε τι προπολογισμό θα χρειαστεί. Αν είμαστε αισιόδοξοι και τα κράτη-μέλη αποφασίσουν του χρόνου να επανακαταστήσουν μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, εναπόκειται στην αρμόδια για τον προπολογισμό αρχή να εξασφαλίσει του απαραίτητου πόρου για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τον αριθμό που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο. Πάντως, γι' αυτό δεν χρειάζεται να συστήσουμε ειδικό πρόγραμμα ή ταμείο. Το ΑΜΙΦ, το Ταμείο Σύλλου Μετανάστευσης και Ένταξης, είναι αρκετό προς το παρόν. Επίσης, το Ταμείο Ασύλου ε, έχει αυτό το εφάπαξ ποσό που πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Τώρα τι κάνουν τα κράτη-μέλη με το ποσό αυτό, δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι, ο, ο όρος είναι να έχει φτάσει ο ενδιαφερόμενος ε, στο κράτος. Να υπάρχει δηλαδή η παρουσία του, η προσωπική, δεν αρκεί η συμφωνία επανεγκατάστασης για να λάβει το κράτος τις 10.000. Επίση, επί της ουσίας, πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω το θέμα τη αιρεσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η επαναγκατάσταση είναι ίσω ένα από τα μελλοντικά μα εργαλεία που θα χρησιμοποιούμε και στι σχέσει μα με τρίτες χώρε σε θέματα μετανάστευση. Πάντω, τονίζω αυτό που είπα και στην αρχή. Δεν θα έχουμε επανεγκατάσταση μόνο για χώρες που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Δεν είναι εκ των ονουκάνευ υπόθεση, ούτε θα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχέδιο θα εκτιμάται περιπτωσιολογικά ανάλογα από τη χώρα, από τις προτεραιότητές μας. Οπότε για συγκεκριμένα σχέδια επανεγκατάστασης αυτά τα θέματα μπορούν να μείνουν κατά μέρο τελείω. Πάντως θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε σε θέση να το χρησιμοποιήσουμε όπου δει και όταν καθορίζουμε και τις μελλοντικές μας προτεραιότητες. Τώρα, στα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Οικογενειακή επανένωση. Μπορεί να είναι νομικό το θέμα. Το θέμα των οικογενειακών δεσμών που προτείνουμε να καλύψει η επανεγκατάσταση δεν ταυτίζεται με τη δυνατότητα που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την οικογενειακή επανένωση. Η δική μας πρόταση είναι ευρύτερη. Δεν ταυτίζεται, επαναλαμβάνω. Γιατί έχουμε πρόσωπα που χρήζουν προστασία σε τρίτη χώρα και μπορεί να έχουν δεσμούς οικογενειακούς, αλλά να μην εμπίπτουν στο, στην κοινωτική νομοθεσία, αλλά να εμπίπτουν στο πλαίσιο της επανεγκατάστασης και να είναι επιλέξιμα με αυτό. Ή μερικοί είναι επιλέξιμοι και με, και με το πρόγραμμα επανεγκατάσταση και με το κοινοτικό αντίστοιχο δίκαιο. Πάντως, με την επανεγκατάσταση, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνοπτική διαδικασία, ίσως είναι ταχύτερη οδός προς την οικογενειακή επανένωση, αλλά όχι πάντα, εξαρτάται από τις συνθήκες. Τώρα για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Είπατε γιατί προτείναμε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Μα γιατί κρίναμε ότι είναι σκοπιμότερο για να καλύψουμε και του εσωτερικά εκτοπιστέντε σε ορισμένε περιπτώσει. Γιατί έχουμε πληθυσμού εκτοπιστέντε εντό του Ιράκ, για παράδειγμα, ευάλωτε ομάδε που έχουν παραμείνει ε, στο, στα όρια μια εθνική επικράτεια και με βάση το ισχύον σύστημα δεν θα ήταν επιλέξει. Με βάση το νέο πρόγραμμα επανακατάσταση θα είναι. Επίσης, άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΥΠΑ της αρμοστίας, αλλά είναι κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτα. Γι' αυτό διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή για να καλύψουμε όλους τους πρόσφυγες για τους οποίους στις χώρες προέλευσής τους δεν υπάρχουν βιώσιμες λύσεις. Γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή του σχεδίου επανεγκατάστασης. Επίσης, αποκλείσαμε αποκλείουμε ένα υποψήφιο που έχει απορρίψει ένα κράτος. Και αυτό είναι θέμα της εναρμόνισης που επιδιώκουμε, γιατί θέλουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μια ευρωπαϊκή διαδικασία. Γι' αυτό, αν κάποιος θέλει να έρθει στην Ευρώπη για σύντομο διάστημα και απορρίπτεται η αίτηση για βραχυπρόθεσμη θεώρηση σε ένα κράτο, δεν θα πρέπει να μπορεί να λάβει τη βίζα από την όμορφη σε ένα άλλο κράτο. Το ίδιο ισχύει για την επανεγκατάσταση. Αν απορριφθεί η αίτηση σε ένα κράτο, είναι σαν να ε, απορρίπτεται σε όλα, γιατί σε όλα τα κράτη ισχύουν οι ίδιε διαδικασίε και τα ίδια κριτήρια. Άρα και η ίδια έκβαση, το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όχι άθροισμα εθνικών. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων γνωρίζετε ότι πολλά κράτη-μέλη μπορούν ε, και μάλλον θα συνεχίσουν για την αποτίμηση κάθε ψηφίου σε επανακατάσταση, θα επαφίονται στην, στην υπατηρμοστία του ΙΕ. Και αυτό θα συνεχιστεί. Γιατί μπορεί κάτι, κάποια κατημέλη να έχουν διαφορετικέ απόψει για το τι θέλουν να κάνουν και εφόσον υπάρχουν ε, διαφορετικέ απόψει μεταξύ του και με το επανεργοστήριο, θα θέλουν να το λύνουν μόνοι του. Για κάθε χώρα που συμφωνεί ε, με την επανεγκατάσταση μπορεί παρόλα αυτά να υπάρχει διαφορετική αποτίμηση από την υποτερμοστία. Οπότε καλό είναι να έχουμε κάποια ευελιξία. Επίση, είμαστε ανοιχτή δυνατότητα να ε, υπολογίζουμε και στην ΙΑΣΟ και στον Μελλοντικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Α, ακόμη, βέβαια, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί τρίτε χώρε δεν είναι ακόμη πολλέ στον αριθμό, αλλά θα μπορούσε αυτό ο οργανισμό να εξυπηρετήσει τα κάτι μελη να α, χειριστούν τη διαδικασία επανεγκατάσταση. Κάτι ακόμη, και είμαι σίγουρο ότι έχω χάσει κάποιε ερωτήσει. Κάτι ακόμη, ποια είναι η σχέση με τα διεθνή προγράμματα, συμπληρωματικά ή εναρμονίζοντα ή στο περιθώριο. Από τη δική μας την ε, πλευρά ελπίζουμε ότι είναι θέμα συμπληρωματικότητας πρώτα απ' όλα. Από την άλλη δεν θα μας πείραζε για να είμαι ειλικρινής από πολιτική σκοπιά, εάν σταδιακά μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έφτασε ο καιρός να πούμε στα κρατημέλη ότι δεν επιτρέπονται τεχνικά τους προγράμματα. Δεν το κάνουμε αυτό. Όμως, αν ε, καλύτερο κόσμο, με μια προοπτική ορισμένων ετών, θα θέλαμε να υπάρχει μια κατάσταση όπου το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανακατάσταση να ε, έχει δημιουργηθεί και τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτά που θέλουν θέλουν ε, ε, για την επανακατάσταση επιπλέον από το πρόγραμμα αυτό, εφόσον το επιθυμούν. Θα μπορούσε να είναι μια μελλοντική εξέλιξη. Ε, με συγχωρείτε για οποιαδήποτε ερώτηση ξέχασα, αλλά βεβαίω είμαστε στην διαρκή διάθεση τη Επιτροπή σα, εφόσον θέλετε να απαντήσω και σε πράγματα που έμειναν απάντητα. Okay, thank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 Είστε έτοιμες και έτοιμοι συνάδελφοι και ιδίω όσοι έχετε εγερθεί και επιθυμείτε να αποχωρήσετε. Είμαστε έτοιμοι και ο διευθυντής του EMCDDA είναι ε, έτοιμος και αυτός να αρχίσει. Παρακαλώ θα μιλήσει όχι πάνω από 10 λεπτά και ετοιμάστε ερωτήσεις εφόσον έχετε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι και πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με, που με ε, προσκαλέσατε να σας παρουσιάσω την έκθεσή μας, να σας ευχαριστήσω και για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη που προσφέρει η Επιτροπή σας στο έργο του οργανισμού μας. Σας ευχαριστώ και για την υποστήριξή σας στην υπερψήφιση του προϋπολογισμού, καθώς και για την υπερψήφιση των τροπολογιών που Επιτροπή σας και τέλος την πολύ ενδιαφέρουσα και δυναμική ε, ε, ε, επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής σας τον περασμένο Ιούλιο. Θα σας παρουσιάσω σύντομα λίγες γενικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Εκθέσεως για τα Ναρκωτικά για το 2016 και θα σας δώσω και κάποιες νοπές πληροφορίες σχετικά με την πορεία του προγράμματος του οργανισμού και ένα τελευταίο σημαντικό σχόλιο θα αναφέρεται στην πρόταση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του κανονισμού μας. Θα ήθελα πρώτα να βάλω ένα πλαίσιο για την έκθεση και να σας δώσω μια οπτική. Πρόκειται για ένα reporting package που ε, συνδυάζει διάφορες πηγές πληροφοριών και την έκθεση που ε, καλύπτει τα τελευταία 10 χρόνια και για όσες και όσους παρακολουθείτε τακτικά τις δημοσίευσεις μας ίσως ορισμένες φορές να αισθανθείτε κάποια σύγχυση αν ήταν δηλαδή έκθεση για την αγορά των ναρκωτικών αν ήταν ε, κάποιο άλλο ε, θέμα, δηλαδή ποιο είναι ο λόγος που βγαίνουν όλες αυτές οι δημοσίευσεις. Αυτή η Drug Market Report που σας παρουσίασα πριν από το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντική. Η ειδική έκθεση που δείχνει με λεπτομέρεια την εξέλιξη της αγοράς ναρκωτικών και την εκδίδουμε ανατριετία. Η έκθεση τάσεων, Trends Report, στην βάση των αναλύσεων που κάνουμε για την τελευταία δεκαετία είναι αυτή που σας υποβάλλω σήμερα και συμπληρώνεται φέτος με δύο ή τρεις άλλες σημαντικές εκθέσεις. Η πρώτη δημοσίευση του κέντρου για, το, για την αγορά ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου. Τον Ιούλιο ξεκινήσαμε μια νέα δημοσίευση για τις πρόσφατες εξελίξεις για την χρήση ναρκωτικών και την υπατήτη ΔΑΓΑΜΑ και τέλος η MCDDA μετά από αίτημα των χωρών μελών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, που ζητήθηκε να σχολιάσει την έκθεση, την μελέτη μάλλον ΕΣΠΑΤ που ήταν η τελευταία πιο πρόσφατη δηλαδή έκθεση για τα σχολεία και κάποια να πούμε πιο σημαντικά θέματα είναι πολύ πλούσια η έκθεση, δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο σήμερα θα σας αναφέρω μερικά από τα πιο σημαντικά σε ό,τι αφορά τη χρήση ναρκωτικών υπάρχουν μικρές αλλαγέ στις τάσεις με την έννοια ότι βλέπουμε να επιβεβαιώνεται μια αύξηση της χρήσης του έκσταση. Ε, υπάρχουν προβλήματα και σε σχέση με τις αμφεταμίνες που επίσης αυξάνεται η χρήση τους στην Ευρώπη και των συνθετικών οπιοειδών. Και μια μέτρια αύξηση των ε, κοινή χρήσεως ναρκωτικών. Θα επανέλθω σε αυτά και πρέπει να τονίσω ότι η καθαρότητα των χαπιών δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε 10-20 χρόνια πριν. Και αυτά οδηγούν σε υπερβολικές δόσεις, σε προβλήματα ε, υγείας και βεβαίως αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν γίνεται, ε, όταν γίνεται συχνή χρήση. Για την κάναβη τώρα υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Βλέπουμε μια αύξηση και σε αυτούς που ζητούν επιζητούν θεραπεία γιατί ε, λόγω προβληματικής χρήσης. Ό,τι αφορά τώρα την αγορά της κάναβης, έχω και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που λέει ότι ένα από τα ζητήματα που ε, είχαμε τελευταία είναι ότι η συγκέντρωση της κάναβης αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα άλλη ουσία που περιλαμβάνεται, περιλαμβάνει η, η στην κάναβη μειώνεται. Τώρα δεν έχει τόση σημασία. Το THC είναι η ε, περιεκτικότητας και, και αυτό έχει ε, σημαντικά ε, ψυχολογικά, σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Άρα μπορούμε να αναμένουμε ότι θα υπάρξει αύξηση, αύξηση της τοξικότητας και των κινδύνων και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν μιλούμε για πρόληψη ή για θεραπεία χρηστών καναβής, τα οποία ήδη εξακολουθούν να είναι σημαντικό πρόβλημα. Κάτι που προκαλεί αύξηση ανησυχία είναι τα συνθετικά οπιοειδή, που περιλαμβάνουν όχι όμως μόνο τις φεταμίνες. Για να εξηγήσω τι εννοώ, στη Νέα Υόρκη ως μέλος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος της εβδομάδας εκείνας, εκείνης είναι διαφορετική στις ΗΠΑ. Οι φεταμίνες είναι πολύ σημαντικές και έχουν αρχίσει και στι ΗΠΑ δηλαδή και έχουν αρχίσει, έχει αρχίσει να αυξάνει τη χρήση του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα θετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν υπάρχουν νέε θεραπείε για την υπατήτητα Γ. Γιατί είναι σημαντικό να μιλήσει κανεί για την υπατήτητα Γ. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν διαφορές μεταξύ χωρών. Όμως, ο αριθμός χρηστών ναρκωτικών είναι μεταξύ 30 και 80% που παθαίνουν υπατήτητα γάμα. Και δεν υπάρχει θεραπεία για τα πρόσωπα αυτά. 20 με 25% θα καταλήξουν τουλάχιστον σε κύρωση και 20% θα, θα καταλήξουν και με καρκίνο του ύπατος, κάτι το οποίο σημαίνει ένα βάρος και για την κοινωνία, τη συλλογικότητα και τα ε, κρατικά συστήματα ασφαλίσεων. Υπάρχει τώρα θεραπεία πρέπει βεβαίω να αναλυθεί το κόστος αυτής της θεραπείας και σας ενημερώνω ότι το κόστος των θεραπείων αυτών έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Για πρώτη φορά όμως υπάρχει πραγματική δυνατότητα οριστικής θεραπείας της ασθένειας. Ολίγα σχόλια για την πρόοδο των δραστηριοτήτων του οργανισμού, γιατί ο χρόνος περνά γρήγορα. Θα θυμάστε ότι στις 10 Σεπτεμβρίου πέρσι εκλέχθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο MCDDA ε, ως ο νέος διευθυντής και είχα το προνόμιο να είμαι παρόν σε ακρόαση την αμέσως επόμενη εβδομάδα και παρουσίασα σε εσά κύριε Πρόεδρε και σε εσά κυρίε και κύριοι το πρόγραμμά μου για τον οργανισμό. Ευχαρίστω σας αναφέρω ότι εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα όπως σχεδιάστηκε και ανακοινώθηκε με σημαντική προτεραιότητα να ενισχύσουμε την απόδοση του οργανισμού. Με την έννοια αυτή έχουμε ενισχύσει και τη συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Ελέγχων που γνωρίζω ότι είναι προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα από τα τελευταία συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λάβαμε ήταν η δήλωση συμφερόντων όλων των μελών του, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής μας Επιτροπής. Και αποφάσισα και εγώ να δημοσιεύσω την δήλωση συμφερόντων μου, παρόλο που για, τον, ε, για τους διευθυντές οργανισμών δεν είναι υποχρεωτική εκ του καταστατικού. Βρισκόμαστε λοιπόν στη, σε σωστή πορεία. Ελπίζω ότι το πρόγραμμά μας θα εγκριθεί από το Managing Board τον Δεκέμβριο Ήδη τον Ιούνιο ήταν πολύ θετικό το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δέχθηκε επίσης και την ε, πολιτική για την πρόληψη απατών και τέλος δύο νέες δραστηριότητες πρώτον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου όλα τα μέλη της Επιτροπής σας και του Κοινοβουλίου θα λάβουν πρόκληση, πρόσκληση συγγνώμη, για να συμμετάσχουν σε ένα νέο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για την κάναβη και τη χρήση της ανά τον κόσμο. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και είναι δύσκολο καμιά φορά να καταλήξει κανείς που βρίσκονται τα πραγματικά γεγονότα για την κειμενική πληροφόρηση και πού είναι κάποιοι ίσως πολιτικοί στόχοι. Και ένας από τους ρόλους του οργανισμού μας είναι να σας προσφέρουμε αντικειμενική ενημέρωση για να καλυφθεί το κενό, για όσους από εσά το χρειάζεστε. Το EMCTDA για το 2017 θα είναι επικεφαλής του δικτύου οργανισμών ε, εσωτερικών και δικαιοσύνης. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της για την αναθεώρηση του κανονισμού του EMCTDA, θέμα για το οποίο η δική σας Επιτροπή πάντοτε έχει το οποίο πάντοτε έχει προσέξει η δική σα Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι ακόμα και αν η διαδικασία άρχισε προτριετίας και κινήθηκε αργά και δύσκολα σε ορισμένε φάσεις, θέλω να πω ότι για την πρόταση αυτή υπήρξε στενότατη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οργανισμού μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την συνεργασία αυτή. Υποστηρίζουμε την πρόταση περιορισμένης αναθεώρησης του κανονισμού μας, γνωρίζουμε και έχουμε και σχετικές συζητήσεις στη διάρκεια της συναντήσεως της Επιτροπής σας, ΛΥΜΠΕ, στο EMCDDA. Υπάρχουν κάποιες ιδέες και κάποιες ερωτήσεις για μια μελλοντική ενδεχόμενη αναθεώρηση της συνολικής εντολής του οργανισμού. Συμφωνούμε όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρώτα χρειάζεται να στερεώσουμε και να μην χάσουμε την εργασία που έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα από τον EMCDDA και να διαθέσουμε και χρόνο σε αυτούς να δούμε ποια είναι και η εξωτερική αξιολόγηση του έργου του EMCDDA που θα γίνει πια το 2018. Σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και πάλι. Γνωρίζω ότι η πρόταση για την αύξηση του προϋπολογισμού είναι σχετικά περιορισμένη. Πρώτα-πρώτα βέβαια πρέπει να είμαστε λογικοί. Μέχρι το 2020 θα αρκεστούμε στα όσα μας προσφέρετε και σας ευχαριστούμε εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Έχουμε όμως χρόνο ακόμη γι' αυτό. Ας επιτύχουμε πρώτα την αναθεώρηση της εντολής και ας συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι καταβάλουμε προσπάθεια για την διαρκή βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού μας. Και εάν χρειαστεί θα ζητήσουμε και έξτρα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Α, βλέπω ότι ο κύριος Ντεπρέ φεύγει. Άρα αφού φεύγει ο κύριος Ντεπρέ, να μην, ίσως να μην συζητηθεί το δημοσιονομικό θέμα. Συνάδελφοι, πριν να προχωρήσουμε στη συζήτηση, να σα ευχαριστήσω για την παρουσίασή σα. Το ίδιο και συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα τη ουσία. Η αντιπροσωπεία μα τον ε, Ιούλιο νομίζω ότι μπορεί να ασχοληθεί με τα επιμέρους θέματα. Όποιος ενδιαφέρεται για αυτά είναι θέματα τα οποία ε, μας ενδιαφέρουν και δεν θέλουμε απλώς να διαφημίσουμε το δικό μας έργο, αλλά πραγματικά συνεισφέρεται σε πολλούς τομείς σε αυτά που μας απασχολούν. Θέλουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έμειναν για να ακούσουν την παρουσίαση. Ευχαριστώ εσάς και όλους, και όλους τους συνεργάτες για τη δουλειά σας. Ε, αρχίζουμε τις ερωτήσεις τώρα με τον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κούστελ, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση και την ποιότητα με την οποία διευθύνεται το κέντρο αυτό. Η Πορτογαλία, η Πορτογαλία ήταν πρωτοπόρος ε, ξεκινήσαμε να αντιμετωπίζουμε την τοξικομανία και τις επιπτώσεις της ε, από τους πρώτους μεταξύ άλλων χωρών. Με όσα μας είπατε βλέπουμε δύο δεδομένα τα οποία φαίνονται κάπως αντιφατικά και θα ήθελα την άποψή σας από αυτού. Από τη μια, η διανομή σιριγκών τοποθετείται την Πορτογαλία στις χώρες με τη λιγότερη έκθεση ελέγχουμε με τη μεγαλύτερη έκθεση ελέγχουμε κατά λιγότερα ποσοστά ε, AIDS, διάδοσης μάλλον του ιού HIV. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Μιλάμε για στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι ζωτική σημασία για την ποιότητα των αποφάσεων που πρέπει να λάβουμε και βάσει της εξαιρετικής μελέτης που μας έχετε κάνει. Ε, Επίση, πολλέ φορέ στι μελέτε μα διαπιστώνουμε ότι απουσιάζουν δεδομένα από κάποια κράτη-μέλη. Κατά την άποψή σα, τι μέτρα θα έπρεπε και μπορούν να ληφθούν ώστε το κέντρο να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση, καλύτερη πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κάρλος. Η Άννα Γκόμες. Σας ευχαριστώ, κύριε Χωστέλ. Είναι πολύ καλό να είστε εδώ και είχα τη χαρά να ηγηθώ της αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε το κέντρο τον περασμένο Ιούλιο. Πραγματικά είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή με, την, ε, με το AMC-DDA. Είναι σημαντικό το τι ζωτικό ρόλο έχει ή το κέντρο σα στην, στην συλλογή ειδικών γνώσεων, ώστε και άλλοι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί να έχουμε μια επί τη ουσία ε, και εύστοχη ανάληψη δράση για να προλάβουμε και το ρυθμό των εξελίξεων. Οι χημικές ανακαλύψεις καθημερινά, οι χημικές εξελίξεις έχουν ε, συνέπειες για την κατανάλωση και την αγορά των ναρκωτικών στην Ευρώπη. από αυτήν την έννοια, πραγματικά με θλίβει αυτό που είπατε, ότι θα χρειαστεί ε, πραγματικά συμφωνώ με αυτό που είπατε για την αναθεώρηση του κανονισμού και θα χρειαστεί και ανάλογη δημοσιονομική στήριξη. Το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που χρειάζεται εδώ υπονοεί υψηλών προσόντων εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα πρέπει διαρκώς να είναι σε δράση και να, να συζητούν με τις αρχές επιβολής του νόμου και των άλλων κρατών και των τρίτων χωρών. Και το θυμάμαι γιατί συμμετείχα και σε αυτό. Συμμετείχα στην επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα πέρσι νομίζω όπου αυτό ήταν πραγματικά μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Είναι πολλές οι νέες ουσίες, διαρκώς ανακαλύπτονται και οι συνθετικές το ίδιο από τους συνδυασμούς τους με ψυχοτρόπες ουσίες διαρκώς να κυκλοφορούν στην αγορά. Ε, πολλές φορές έρχονται από την Μέση Ανατολή, το Λίβανο, μέσω λιβάνου από την Κίνα και η σύσταση κάποια φορά, κάποιες φορές είναι εντελώ άγνωστη στον υπόλοιπο κόσμο. Καλό είναι λοιπόν που το κέντρο μπορεί να κάνει αυτό του είδους την καταγραφή στοιχείων. Επίσης, γι' αυτό χρειάζεται και πόρους. Και Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα χρειαστεί ε, μεταξύ μα συνεργασία και συντονισμό για να μπορούμε από κοινού να αναχαιτήσουμε τι αρνητικέ επιπτώσει από τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα. Από ό,τι είδαμε με την επίσκεψή μα εκεί, οι Κινέζοι παραδέχτηκαν ότι εντάξει, τη γνωρίζουμε την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε για τίποτα γιατί αυτά τα προϊόντα έτσι καλλιώ εξάγονται. Δεν μα αφορούν εσωτερικώ ω του καταναλωτέ του. Αυτή ήταν η στάση του και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει διωγγώσει εκθετικά την, ε, τις διαστάσεις του φαινομένου. Απλώς να θυμίσω ότι στην επίσκεψη στη Λισαβόνα νομίζω έμαθα και κάτι το οποίο αναφέρεται φέτος σε όλες τις συζητήσει Είναι ιδιαίτερη σημασία για, το συσχετισμό που κάνατε με τις τρίτες χώρες και όλο ιδιαίτερο στην Ιορδανία. Όταν έγινε η... όταν εντοπίστηκε το φορτίο ενός ε, σκάφους ενός πληρώματος που υποτίθεται ότι το διακινούσαν οι μέλη του ISIS. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν οι πληροφορίες που συλλέγεται, όχι μόνο για τα θέματα ελέγχου και παρακολούθησης στον τομέα της κατανάλωσης ναρκωτικών και τοξικομανίας και έθισμου, αλλά και για άλλους τομείς της δραστηριότητάς μας, όπου είναι πολύ σημαντική ούτως ή άλλως για την ασφάλειά μας συνολικότερα. Ευχαριστούμε η Μαϊτέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και να συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Αισθανίζομαι σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα σχόλιά τους. Με προβληματίζει και με ανησυχεί που πολλές χώρες δεν έχουν δώσει ακόμη τα στοιχεία τους ε, για να δημιουργήσουμε δείκτες, γιατί μας χρειάζονται δείκτες και θέλουμε να παραμείνει ε, το κέντρο παρακολούθηση, το κέντρο αριστεία. Μερικέ φορέ το φθηνό το πληρώνουμε ακριβά, ενώ το ακριβό μα βγαίνει φθηνά. Και νομίζω ότι επειδή μιλούμε για του νέου, ε, μα ενδιαφέρει να δουλέψουμε με ενθουσιασμό, ζήλο και αυτό νομίζω ότι είναι και το σήμα κατά τεθέν, αυτός ο ζήλος και ενθουσιασμός του κέντρου παρακολούθησης ε, και αυτό το στίγμα δώσατε και εσείς με τη δική σας θητεία. Φυσικά θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους δείκτες και τους, τις, ε, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και φυσικά χρειάζεται πόρους γιατί χωρίς πόρους οι ίδιες αυτές εκθέσεις ε, θα μετατραπούν ε, σε κάτι τετριμένο και δεν θα προκαλούν ενδιαφέρον. Θέλουμε να παραμείνει το κέντρο παρακολούθηση ναρκωτικών και τοξικομανίας ω κέντρο αριστείας. Επίση, είναι σημαντικό να έχετε και εσωτερικού ελέγχου Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για το δικό σας οργανισμό, αλλά και για άλλους ε, ε, κρατικούς φορείς και διεθνείς. Αυτά και πείτε μας ε, τι περιεχόμενο να δώσουμε στις τροπολογίες που θα καταθέσουμε και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του κέντρου σας. Ευχαριστώ, κύριο Κοράου. Yes, thank you, sir. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χόρτελ για την παρουσίασή σα. Ήμουν και εγώ ένα από αυτού που ταξίδεψαν τον Ιούλιο στη Λισαβόνα για να σα επισκεφτώ και είχα τη χαρά να συζητήσω για την έκθεση αυτή μαζί σα και με του συνεργάτε σα και για τόσα κάνει το κέντρο. Συμφωνώ απολύτω με όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους για την ανάγκη να υπάρχουν ε, σωστές πληροφορίες με τους κατάλληλους δείκτε και, και να διατηρήσετε την αριστεία σας για να μπορούμε και εμείς να εκπονήσουμε σωστά τις πολιτικές μας. Όμως κάτι που διαφαίνεται ξεκάθαρα από την έκθεση είναι ότι ένα τεράστιο μερίδιο της αγοράς το καταλαμβάνει η κάναβης. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ξανά το πώς σχεδιάζουμε τις πολιτικές μας ή να συζητάμε σε αυτό το κοινοβούλιο για την κάναβη, για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που έχει αποτύχει ως τώρα. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε να ξεκινήσει η συζήτηση για αλλαγή των πολιτικών μας ε, για την κάναβη και τα υπιότερα ναρκωτικά. Τα πιο ε, ανώδυνα ναρκωτικά όπως θεωρούνται. Να δούμε μήπως είναι διαφορετικές οι συνέπειε τους από ό,τι θυμόμαστε στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα είναι Βλέπουμε προβληματικά τα στοιχεία εδώ στην έκθεση και υπάρχουν διαφορετικά είδη της κάναβης που δύσκολο είναι να καταγραφούν. Συνάδελφε, κανείς άλλος, πριν δώσω το λόγο στον Διευθυντή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Απαντήστε αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις ε, γιατί μερικές φορές αλληλοεπικαλύπτονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τα μέλη της Επιτροπής σας που ήρθαν και σήμερα, αλλά και συμμετείχαν στην αποστολή στο κέντρο στη Λισαβόνα, γιατί έτσι είχαμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε την προστιθέμενη αξία του έργου μας και να ενισχύσουμε αυτό το συνδέσμο μεταξύ της ε, παραγωγής πληροφοριών και τη στήριξη των δράσεων, δηλαδή τη στήριξης της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι ε, περισσότερες ερωτήσεις αναφέρθηκαν στους δείκτες και στην έλλειψη πληροφοριών που έχουμε από τα κράτη-μέλη. Εδώ έχουμε διαφορετικές ε, καταστάσεις. Μερικοί δείκτες συγκεντρώνονται περιοδικά για παράδειγμα, δημοσκοπήσεις στο γενικό πληθυσμό, οι μελέτες για το γενικό πληθυσμό. Και για δεδομένο χρόνο ε, μας έλειπαν στοιχεία από μία-δύο χρόνες, γιατί η περιοδικότητα ή ο κύκλος τέτοιης συλλογή στοιχείων δεν συμπίπτει με τη χρονιά της εκπόνησης της έκθεσης. Ή έχει αλλάξει ο κύκλος μερικές φορές. Πάντως, ένα σημαντικό και ανησυχητικό σε ορισμένες χώρες θέμα είναι η γενική κατάσταση του εθνικού προϋπολογισμού, όχι μόνο για τη δημόσια υγεία, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Και αυτό είναι ένα από τα ε, δυνάμει ενισχυτικά θέματα. Ένα άλλο θέμα αφορά ε, την ποιότητα των στοιχείων, την κάλυψη των στοιχείων και μεθοδολογικά θέματα. Εκεί έχουμε κάποιους περιορισμούς. Και ένα τρίτο ζήτημα, ίσως από τεχνική άποψη μία μελέτη είναι καλή ως προς την περιγραφή της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, αλλά για τεχνικούς λόγους, επειδή δεν χρησιμοποιείται η ίδια μεθοδολογία, δεν είναι συγκρίσιμη με άλλες μελέτες άλλων χωρών που χρησιμοποιούν άλλη μεθοδολογία. Επίσης, ό,τι αφορά τους δείκτες ε, προσφοράς. Πριν από λίγα χρόνια το κέντρο μας ανέλαβε εντολή από την Επιτροπή και το Συμβούλιο εκτιμήσει από κοινού με τη Europol την κατάσταση και να υποβάλει πρόταση για τη βελτίωση και την εδραίωση των συγκεκριμένων δικτών. Είχαμε όμως δύο διαφορετικές θέσεις. Καταρχήν είχαμε την κατάσταση πριν την μείζωνα χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τότε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη επιθυμούσαν μια φιλόδοξη πρόταση και πρώτης κρίσης. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ε, σκεφτόταν ακόμη και την πιθανότητα αύξηση του σχετικού προπολογισμού. Στο μεταξύ όμως μεσολάβησε η σοβαρότατη αυτή η οικονομική κρίση και στην τελική διάσκεψη για, την, ε, για τους δείκτες η θέση των κρατών μελών ήταν θέλουμε μεν πρόταση αλλά δεν έχουμε ούτε ένα ε, δεν θέλουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον να ξοδεύσουμε σε εθνικό επίπεδο και ούτε να αυξήσουμε και τον ευρωπαϊκό σχετικό προϋπολογισμό. Οπότε θέλουμε να βελτιώσουμε το έργο για τους δείκτες, αλλά γι' αυτό επαφιόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο έργο του προσωπικού του Κέντρου Παρακολούθησης και σε κάποιους ιδρύκους εμπειρογνώμονες. Οπότε ο ρυθμός βελτίωσης και εξέλιξης του έργου επί των δικτών δεν είναι τόσο γρήγορος όσο ελπίζαμε αρχικά. Και τι κάνουμε γι' αυτό. Εμείς στην προσέγγιση μας έχουμε ε, τρία-τέσσερα επίπεδα. Καταρχήν, ε, στήριξη, μεθοδολογική, ακόμη και κατάρτιση στα κράτη-μέλη για να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα. Δεύτερον, διάλογος. Για παράδειγμα, τον Μάιο ε, πήγα μετά από επίσημη πρόσκληση σε ένα κράτος μέλος για να συζητήσουμε το θέμα της μη διαθεσιμότητας προς το Κέντρο Παρακολούθησης των Εθνικών Στοιχείων για τις Κατασχέσεις. Έχουμε ξεκινήσει έναν καλό διάλογο και θα έχουμε και τον επόμενο μήνα μια τεχνική συνάντηση για να δούμε αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Άλλο παράδειγμα, η Σουηδία που προσκάλεσε το κέντρο παρακολούθησης για να τη βοηθήσουμε να βελτιώσει και να καταλάβει καλύτερα ε, το πώς λειτουργούν οι δείκτες της σημότητας λόγω ναρκωτικών ε, στη χώρα. Οπότε έχουμε και με τη Σουηδία τέτοια συνεργασία. Επίσης, αλλάξαμε την προσέγγισή μας, οπότε δεν μπορούμε να επαναλάβουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τεχνολογίες για τους δείκτες προσφοράς με αυτούς που χρησιμοποιούσαμε για τους βασικούς επιδημιολογικούς δείκτες, γιατί αυτοί ξεκίνησαν πριν από 25 χρόνια και τότε δεν είχαμε αρκετά κονδύλια τότε σε, ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε προσαρμόσαμε το έργο και τη μεθοδολογία μας, λαμβάνοντα υπόψη και αυτό τον περιορισμό και τέλος, πριν φτάσω στην απάντηση προς τον κύριο Κοράο, εγώ ως διευθυντής του Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας πιστεύω ότι αν θέλουμε να χάσουμε τη στήριξη από τις επενδύσεις των κρατών μελών θα πρέπει να ενισχύσουμε και να κάνουμε ε, πιο ορατή, να προβάλλουμε καλύτερα την προστιθέμενη αξία του κέντρου μας στα κράτη-μέλη. Και αυτή είναι η βασική προτεραιότητα της ε, καινούργιας μας στρατηγικής. Και ως προς την ερώτηση του κύριου Κοράου, και του κυρίου Κοέλιο. Να ξεκινήσω από την ερώτηση του κυρίου Κοέλιο. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Δεν θα κάνω πιθανολογίες τώρα, θα ρωτήσω το, τους συνεργάτες μου. Πάντως, ε, τα στοιχεία για τον ιό του AIDS στην Πορτογαλία ε, και το υψηλό όπως το επιπολεσμό ήταν ιστορικά στοιχεία. Δηλαδή, η συμπεριφορά κινδύνου εξακολουθεί να είναι έντονη. Θα σας στείλω πάντως και γραπτή απάντηση και είναι σημαντικό να έχουμε προγράμματα διανομής ειρηνικών γιατί το θέμα είναι συναφές με την επικίνδυνη συμπεριφορά. Όταν βελτιωθεί αυτή η επικίνδυνη συμπεριφορά μεταξύ των χριστών, αλλά ακόμη και όταν ε, ε, ε βελτιώνεται η επικίνδυνη συμπεριφορά λόγω διανομής, όλα αυτά τα κρούσματα οροθετικών ήταν υψηλά. Πάντως θα το διερευνήσω και θα σα στείλω γραπτή απάντηση. Προ τον κύριο Κοράο, φυσικά δεν ήταν εύκολη ερώτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θεωρώ σημαντικό όλοι οι οργανισμοί να σα δίνουν ουδέτερες αντικειμενικές αμερόληπτες πληροφορίες για το τι συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές του κόσμου, στι Ηνωμένες για παράδειγμα και άλλου. Γι' αυτό και τον Οκτώβριο θα έχουμε το νέο ειδικό σύστημα για την προειδοποίηση. Για το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων τώρα, όπως ε, συζητήσαμε και τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της διάσκεψης, αν έχουμε 15 ή 20 χώρες ε, ε, που έχουν ε, νομιμοποιήσει και παράγουν ε, νόμιμα κάναβη θα έχει κάτι τέτοιο ε, αντίκτυπο και στην πολιτική συζήτηση και στην εξέταση των πολιτικών επιλογών. Όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σίγουρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρο τη Κολομβίας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να τιμωρήσει τους αγρότες που καλλιεργούν μαριχουάνα στην Κολομβία, ενώ η καλλιέργεια μαριχουάνας είναι νόημη σε μερικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση λοιπόν από αυτό είναι σημαντική και θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε ρόλο, ακόμη καλύτερο μάλιστα από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, για να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και να σας βοηθάμε στη διεξαγωγή της συζήτησης. Έκανα ένα μικρό λάθος. Θα έπρεπε να είχα δώσει το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πριν από εσά. Λυπούμε πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο γιατί δεν έχει αγαλθεί ακόμη η κυρία Μακοβέη που είναι αρμοδία για το επόμενο θέμα. Αν θέλετε λοιπόν μπορούμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε να κάνετε, ε, κυρία εκπρόσωπη της Επιτροπής, μια σύντομη ε, τοποθέτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ευχαριστώ να παρέμβω τώρα και ευχαριστώ τον Διευθυντή του Οργανισμού EMCDDA για την παρέμβασή του, καθώς και την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών για την διοργάνωση της ανταλλαγής απόψεων. Δύο πράγματα έχω να πω. Αφενός, όπως είπε ο Αλέξης, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει στις 29 Αυγούστου νέα πρόταση η οποία θα οδηγήσει στην αλλαγή της νομικής βάσεως για τον οργανισμό για να προβλέπετε και σύστημα έγκυρης προειδοποίησης αλλά και αξιολόγησης κινδύνου που είναι πολύ σημαντικά και για το σύστημά μας MPS είναι τμήμα συμβιβασμού που ε, η Επιτροπή σας θα υποστηρίξει για να λυθούν ορισμένα από μακρού υφιστάμενα προβλήματα για τις αποφάσεις του MPS θα αντιμετωπιστούν με ταχύτητα από την Επιτροπή σας και από το Κοινοβουλίο. Σημαντική διάσταση της προτάσεως είναι η δημοσιονομική πτυχή. Θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά μετά από μία τριετία προτείνει αύξηση της ε, Ευρωπαϊκής Ενωσιακής Επιδότησης για το EMCA για ένα εκατομμύριο δηλαδή για το υπόλοιπο εναπομένων ένα έτος δραστηριότητας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την ε, ε, πίστοση αυτή και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, στην νομοθετική της πτυχή και στη δημοσιονομική της πτυχή. Τώρα η διεθνής διάσταση της πολιτικής για τα ναρκωτικά είναι σημαντικό να έχει δύο σκέλη. αφενό την διεθνή δράση και αφετέρου τη δράση εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με την κυρία Γκόμε για την σημασία της Κίνας που είναι εταίρος μας, ελπίζουμε, για το μέλλον και που θα πρέπει να διεξαχθεί με τη μεγάλη αυτή χώρα ένας ορθός διάλογος για τα ναρκωτικά γίνονται και διαπραγματεύσεις στην Ούγκας. Πολύ δύσκολες συζητήσεις άλλωστε ιδίως για το θέμα της ε, επιβολής της θανατικής ποινή για αδικήματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά. Παρ' όλα αυτά η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα όπως είπα η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξάγει δηλαδή ε, ε, διάλογο μαζί της για τη μετώπιση δυσχερών θεμάτων. τουλάχιστον σε επίπεδο MPS. Γίνεται διάλογος για, τη, για, για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, όχι ακόμα για το MPS. Ευχαριστώ. Και λυπούμε πολύ και πάλι για την παραδρομή προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ και εσάς και το προσωπικό σας. Υπήρχαν και ορισμένα θέματα προπολογισμού, τα οποία ίσως δεν απαντήσαμε ε, με πληρότητα, αλλά αυτό θα χρειαστεί να περιμένει για να γίνει κάποια άλλη φορά. Ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συμβολή σας στην συζήτηση των σημαντικών αυτών θεμάτων. Ευχαριστώ. Τώρα θα προχωρήσουμε στο πρώτο τελευταίο θέμα, υπαριθμόν 6, που είναι η ενίσχυση των ελέγχων στη βάση τραπεζών δεδομένων και για τα εξωτερικά σύνορα. Και η εισηγήτρια είναι η Μάκοβέη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για πρόταση τροποποίησης του κώδικα Schengen για τα σύνορα για να περιληφθεί η υποχρέωση των χωρών μελών να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους στην βάση τραπεζών δεδομένων για υπηκόους τρίτων χωρών και για ανθρώπους οι οποίοι διακινούνται ε, στην βάση του κοινοτικού δικαίου και επομένως για υπηκόους χωρών μελών όταν διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα εφόσον είναι ε, θέμα δημοσίας τάξεως και ασφαλείας. Έχει γίνει, έχουν ε, γίνει οι σχετικοί τεχνικοί διάλογοι Έχουμε τέσσερα βασικά στοιχεία που είναι αμφιλεγόμενα αυτή τη στιγμή και όπου το Συμβούλιο αρνείται να μετακινηθεί από τις θέσεις του και πρόκειται για πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Τα τέσσερα αυτά σημεία για την ε, επιβολή ελέγχων σε χερσαία εναέρια κλπ. σύνορα Υπάρχει κείμενο της Κομισιόν, γίνεται όμως δυνατόν να γίνει, υπάρξουν εξαιρέσεις και στα ενέργεια σύνορα ε, στη βάση του κειμένου της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Το Συμβούλιο δεν θέλει εξαίρεση. Οποτεδήποτε για ενέργεια σύνορα. Γι' αυτό προτείνουν περίοδο εξαμήνου ώστε να εξοπλιστούν τα αεροδρόμια χωρίς άλλες εξαιρέσει. Και μόνο στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Το Συμβούλιο εμένει στη θέση του. Δεύτερο σημείο διαφωνίες λόγοι εξαιρέσεων για στοχευμένους ε, ελέγχους το Συμβούλιο συμφωνεί με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εφαρμόζει στοχευμένους ελέγχους στην βάση πληροφοριών που έχει για άτομα μόνο εάν υπάρχουν εξαιρετικές κυκλοφοριακές ροές ώστε να μην χρειάζονται πλέον, ή μάλλον να μην είναι δυνατόν να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι και να γίνονται μόνο στοχευμένοι έλεγχοι. Το κείμενο που εγκρίθηκε στην ΛΥΜΠΕ για να εφαρμόζουν οι χώρες στοχευμένους ελέγχους όταν διαπιστώνουν ότι οι συστηματικοί ελέγχοι έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις γενικά όχι μόνο στην κυκλοφορία, γενικευμένα σημαίνει σε οποιαδήποτε ε, περίσταση. Είναι αόριστη διατύπωση. Το τρίτο, η διαβούλευση, ο έλεγχος στην βάση τραπεζών δεδομένων. Κείμενο της ΛΥΒΕ, που δεν περιλαμβάνει πλέον σε εθνικές τράπεζες δεδομένων, ενώ το Συμβούλιο ακολουθεί την πρόταση της Κομισιόν και επιμένει να μπουν στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο θα γίνεται η διαβούλευση και οι εθνικές τράπεζες δεδομένων. Και τέλος η καταληκτική ρήτρα στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών εγκρίναμε τροπολογία που λέει ότι ο κανονισμός λύγει μία πενταετία μετά από την θέση ισχύ του. Το Συμβούλιο είναι απολύτως αντίθετο εν προκειμένου. Λόγω των θεμάτων αυτών επιτελέστηκε πολύ λίγη πρόοδος στον ε, πολιτικό τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι έχει οριμάσει ο χρόνος. Χρειάζεται να ελέγξουμε αποτελεσματικότερα τα σύνορά μας. Περισσότερο αποτελεσματικά από ό,τι ποτέ. Ε, σωστό αυτό που λέτε, απαντά ο Πρόεδρος. και μπορείτε να ολοκληρώσετε με, το, με, την, ε, με την άποψη αυτή. Ευχαριστώ, αλλά ίσως έχουν κάτι να πούνε οι συνάδελφοί μου. Ευχαριστώ πολύ. Εκ των σκιωδών. Η κυρία Κουντρίτσκα που είναι η σκιώδη συγγετρία από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέη αλλά και το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Είχαμε πολλές ε, επαφές και συναντήσεις και σε τεχνικό επίπεδο και στον τριμερή διάλογο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανέκυψαν κάποιες διαφορές και τεχνικές και ενοιολογικές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την έννοια των συνόρων ε, με βάση ποιο κριτήριο θα εισάγουμε στοχευμένους κινδύνους τα, τις εθνικές βάσεις δεδομένων, αλλά και το θέμα της ε, ε, εισαγωγής ρητρών λήξης ισχύω, sunset clause. Θα πρέπει να βρούμε συνενετική λύση στο μέτρο του δυνατού, ε, δεδομένων και των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων, γιατί το υπέρτερο αγαθό είναι η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία και η διαφύλαξη των εξωτερικών μας συνόρων. Για μας το ΕΛΚ ε, ζητούμενο είναι η αναζήτηση αποτελεσματικής λύσης για να τεθεί στο συντομότερο δυνατό σε εφαρμογή ο κανονισμός. Αυτό είναι ο στόχος μας και θα συνεργαστούμε για να τον ελοποιήσουμε. Θέλουμε επικοδομητική ανταπόκριση και από το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να καταλήξουμε σε συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μπάρμπαρα. άλλο και όδη κάποιο συνάδελφο που να είναι εδώ. Εάν όχι, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μακοβέη. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ. Μια ακόμα κουβέντα. Συμφωνώ με τη συνάδελφο. Είναι πήγον να βρεθεί λύση στο θέμα. Ήλπιζα να εγκριθεί πριν τις διακοπές. Νομίζω και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να δείξουν κάποια ευελιξία συμπεριλαμβανομένων των ε, συναδέλφων από τις υπόλοιπες ομάδες και ελπίζω να εγκριθεί ο κανονισμός αυτός που είναι πολύ σημαντικός για την προστασία των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την ενημέρωση. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στο σημείο 7. Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Αλλά διερωτώ Κοιτάζοντα τη Μόνικα, τη συντονίστρια μα από το ΕΛΚ, θα αναλάβει εσύ. Α, εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερω. Σημείο 7 λοιπόν. Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Συγητή είναι ο κ. Πάμπρεξ. Δυστυχώ όμω δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε θα τον αντικαταστήσει η συντονίστρια του ΕΛΚ, η κυρία Χόλμαγερ. Ε, μιλάμε για την εξέταση της έκθεσης αυτής και βάσει το άρθρο 200 και μάλλον βάσει το εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου θα αναλάβει το θέμα η Μόνικα, θα περάσει από την, Ολο... πέρασε από την Ολομέλεια τον Ιούλιο και βρισκόμαστε στη διαδικασία της ε, συναπόφασης. Όπως είπα, δεν μπορεί να είναι εδώ ο κ. Πάμπικ σήμερα. Η κ. Χολμάγερ θα μας αναπτύξει το θέμα. Παρακαλώ, Μόνικα, λάβε το λόγο και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πάμπριξ σας απευθύνει χαιρετισμό, δυστυχώς κολλείεται και γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνω εγώ την ε, τιμή και την ευθύνη να σας διαβάσω αυτά που έχει γράψει. Ο εισηγητής λοιπόν ευχαριστεί πρώτα όλους τους και εισηγητές, Συμβούλου, ε, ε, πρόσωπα της γραμματείας καθώς και του γλωσσομαθεί νομικού για την ε, συμβολή του, Όλων τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εμά. Έχουμε όλοι εργαστεί έντονα για να ολοκληρώσουμε έγκαιρα αυτή τη σημαντική νομοθεσία. Στις 6 Εβδόμου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τον κανονισμό για την συνοριοφυλακή, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Όμως η ψήφος αυτή έγινε επικειμένου που είχε συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ των διαπραγματευτών. Συνήθις πρακτική σε περιπτώσεις όπου το εφιστάμενο χρονικό πλαίσιο είναι πολύ σύντομο και δεν επιτρέπει πλήρη έλεγχο. Μετά από την κοινοβουλευτική ψηφοφορία, οι γλωσσομαθείς συνομικοί εξέτασαν το κείμενο για να του δώσουν την τελική ορθή νομοτεχνική μορφή. Ο εισηγητή είναι ικανοποιημένο από την εργασία των γλωσσομαθών νομικών, θεωρεί ότι οι διορθώσεις είναι ορθές και βεβαίω μέσα στο πνεύμα της πολιτικής συμφωνίας που είχε προηγηθεί. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, διαθέσει τις ε, αναγκαίες δυνάμεις καθώς και το απαραίτητο υλικό. Αυτά λέει ο αγαπητός Πάμπριξ που τα συνδυάζει με τις ευχαριστίες του προς όλες και όλους τους συναδέλφους καθώς και προς την γραμματεία της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε για την τόσο ε, καλή επισκόπηση αυτού του τόσο σημαντικού θέματος. Να πω, συνάδελφοι, για να γραφτεί και στα πρακτικά και επειδή έχω κοιτάξει το κείμενο και με όσα είπε και η Μόνικα, Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει από την Επιτροπή μα να, να θεωρήσουμε ότι οι διορθώσεις που υποβλήθηκαν σήμερα, το διορθωτικό δηλαδή είναι ικανοποιητικό και μπορούμε να το στηρίξουμε. Θα ενημερώσω τι ε, υπηρεσίες της Ολομέλειας για τη σημερινή μα συζήτηση. Μετά το διορθωτικό θα περάσει από την Ολομέλεια βάσει του άρθρου 231 παράγραφο 4 και θα εγκριθεί από το Συμβουλίο στι 14 Σεπτεμβρίου, ενώ θα υπογράψουν οι σκιώδει του Στρασβούργο την ίδια ημερομηνία και έπειτα θα δημοσιοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Για να περάσει από την Ολομέλεια, όπως ε, καταλαβαίνετε, την ερχόμενη εβδομάδα βεβαίως, έτσι. Ευχαριστώ πολύ Μόνικα, ευχαριστώ συνάδελφοι. Περιμέναμε αυτή την ανακοίνωση για να ολοκληρώσουμε και με το σημείο 7. point. Πάμε στο σημείο 8, διάφορα. Εάν δεν υπάρχουν διάφορα, οι επόμενε συνεδριάσεις μας, σημείο 9, 12 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα στο Στρασβουργό ακρόαση του υποψήφιου επιτρόπου για την ε, Ένωση Ασφάλειας από το Ηνωμένο Βασίλειο, του κυρίου Τζούλιαν Κίνγκ.